Allora, we can start now. Ciao. Να eh, ξεκινήσουμε λοιπόν. Να πω λίγα λόγια. Πριν να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας. Έγκριση μερίσιας διάταξη. Συμφωνείτε, αν συμφωνείτε, θεωρούμε εγκεκριμένη την ημέρα σε διάταξη. Όσον αφορά τι ανακοινώσει, Έχουμε διερμηνία γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, δανέζικα, ελληνικά, Σπανικά, τσεχικά, εστονικά, ουγγρικά, μαλτέζικα, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Είμαστε και στο διαδίκτυο. Έχουμε web streaming και στείλαμε σε όλους τους συναδέλφους το σημείωμα με τις αποφάσεις των συντονιστών της 18ης Απριλίου και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσει, θεωρούνται εγκεκριμένα πρακτικά. Πριν περάσω στο σημείο 3 και δώσω το λόγο στη Σαμπίνα, την συγγήτρια, θέλω να χαιρετήσω, να κάνω μάλλον μια, δύο, δύο-τρει μάλλον σύντομε ανακοινώσει. Με συγχωρείτε κιόλα, γιατί έχω κρυολογήσει. Λοιπόν, πρώτα, όπω είπα και στου συντονιστέ και το επαναλαμβάνω και στην Επιτροπή, ότι έχω διανύμει όπως έπρεπε την παρέμβαση που έκανε όματι της Επιτροπής όταν προσεκλήσε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτισμού ε, που έγινε την προηγούμενη Τρίτη, πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Περίπου 900 άτομα όλων των χωρών ήταν παρόντα. Πάρα πολύ υψηλή ποιότητα. Έχετε κάποια, κάποιο πρόβλημα με τη διερμηνία, Τερέζα. Στα αγγλικά έχουμε παρεμβολές, θόρυβο. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με παρεμβολές και θόρυβο. Αλλάξατε μικρόφωνο. Καλύτερα, ωραία. Έλεγα λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ στις Βρυξέλλες, Φόρουμ Πολιτισμού, Δευτέρα και Τρίτη 18 και 19 έγινε, συμμετείχα, μίλησα στην εναρκτήρια ομιλία μετά τον Επίτροπο Ναύρατσιτς και με τα χαράς συνάδελφους που δεν μιλήσαμε. Σας λέω λοιπόν ότι δύο σημαντικότατα νέα έχουμε. Πρώτα απ' όλα καταφέραμε σαν Επιτροπή διότι πιστέψτε με ήταν προσωπική προσπάθεια που κατέβαλα και είχα και σημαντική υποστήριξη όμως από τον πρόεδρο Σούλτς καταφέραμε λέγω να έχουμε έγκριση από πλευράς του σχεδίου Γιούνκερ για το 2018 να θεωρηθεί το 2018 Ευρωπαϊκό Έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θεωρήθηκε χαμένη μάχη αλλά κερδίσαμε. Τους επόμενους μήνες λοιπόν ο Επίτροπος Ναύρασιτς θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα εργασιών και βέβαια εγώ ζήτησα από τον Επίτροπο Ναύρασιτς να συμμετάσχουμε σαν Επιτροπή και σαν Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του προγράμματος. Δεύτερο, καλό μαντάτο. Επίσημα ανακοινώθηκε από την ύπατη εκπρόσωπο την κυρία Μογκερίνη η παρουσίαση μιας ανακοινώσεως με θέμα η νέα πολιτική διεθνών σχέσεων, πολιτισμική πολιτική για τις διεθνείς σχέσεις. Άρα η διπλωματία του πολιτισμού, culture diplomacy. Στο Συμβούλιο Υπουργών θα παρουσιαστεί στις 30 και 31 Μαΐου και, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μεγάλη προσοχή που δόθηκε σε αυτό και από την πλευρά μας θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους της Επιτροπής ΑΦΕΤ, Εξωτερικής Πολιτικής, χρειάζεται ε, συνεργασία. Έχουμε τρεις επιτρόπους οι οποίοι θα ε, παρουσιάσουν τις προσπάθειές τους με, υπό την ηγεσία της ύπατης εκπροσώπου. Ενδιαφέρει, ενδιαφέρουσα προσπάθεια. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που συμμετείχαν. Την Helga Truppel ευχαριστώ, διότι από τον, από τον Ιταλό Υπουργό Φραντσεσκίνη παρουσιάστηκε το σχέδιο Task Force για τους ε, του πολιτισμού. Η Ιταλία ήδη έδωσε 30 άτομα για την Task Force. Ε, οι 30 είναι η ειδική μονάδα των αστυνομικών που είναι ειδικευμένη για έργα τέχνη, για την προστασία τη πολιτιστική κληρονομιά και ανάκτηση των έργων τέχνη και 30 είναι αρχαιολόγοι, εμπειρογνώμονε κλπ. Ανταποκρινόμενε στην έκκληση τη Ειρήνα Μπουκόβα τη UNESCO του Εκταλιστικού Συμβουλίου ε, του περασμένου Οκτωβρίου. Πιστεύω ότι όλοι σα σίγουρα θα συμφωνείτε να ευαισθητοποιήσετε τα διάφορα κράτη-μέλη και έτσι αυτό να γίνει ένα πρόγραμμα και μια προσπάθεια όλων των κρατών μελών και δέσμευση. Αλλά εκείνο που μου με ευχαρίστησε ιδιαίτερα το είπατε εκπρόσωπος η κυρία Μογκερίνη ανακοίνωσε ότι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει στον ΟΗΕ αυτό να το κάνει σαν μάχη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι σημαντικό διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε πρώτο αυτό το θέμα της ε, σειράς μέτρων για να μην καταστρέφεται η πολιτιστική κληρονομιά. Ένα από αυτά είναι ειδική ομάδα κρούσης, task force, για τα πολιτιστικά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω άλλα στις ανακοινώσεις, τουλάχιστον για την ώρα. Ορίστε. Α, ναι, μάλιστα. Πριν σας δώσω το λόγο, στο σημείο 3 θα ήθελα να δώσω μάλλον τώρα το λόγο. Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν σας είδα. Ε, κύριε Φίσας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι χτες ακριβώς υπήρξε μία έγινε μία εκδήλωση στη Βαρκελόνη για τον Πλάσιντο Ντομίγκο ήταν 40η επέτειος της πρώτης ε, παράστασης που έδωσε σε αυτό το θέατρο ε, είναι παρόν στο Ευρώπα Nostra και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο ο Πλάσιντο Ντομίνγκο που έχουμε αυτή την εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Κληρονομιάς της Πολιτιστικής. Ήταν πολύ ικανοποιημένο με τις προσπάθειες που έκανε το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτό το τομέα. Μου ζήτησε να διαβάσω τα θετικά του αυτά σχόλια. Στο τέλος Μαΐου θα έχουμε μία εκδήλωση και θα παρουσιαστεί αυτό το πρόγραμμα. Θα είναι παρόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίσας. Σίγουρα ε, ε, πολεμήσαμε για αυτό το αποτέλεσμα. Η Ευρώπα Νόστρα πολέμησε γι' αυτό. Κάναμε πολλές προσπάθειες και ξέρω ότι είχε ανακοινωθεί αυτή η πρωτοβουλία στη Μαδρίτη. Το σημαντικό είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορέσουν να συνεργαστούν και ξέρω ότι και το Συμβούλιο δημιούργησε μια ομάδα προβληματισμού, Reflection Group, από αυτού, οπότε σίγουρα έχουμε σημαντικό έργο μπροστά μας. Για να δώσω το λόγο τώρα στη Σαμπίν Φεράιερ, που είναι η συγγήτρια για την νομοθετική πρόταση όσον αφορά την, ε, τη, μεταφορικότητα. Subito, ε, τη φορητότητα την ευρωπαϊκή ε, των, στοιχείων. Λοιπόν, θεωρώντας ότι είναι περίπλοκο θέμα και θα πρέπει να υποβληθούν τροπολογίες για το θέμα αυτό της φορητότητας. Εκτός μικροφώνου ένα διάλογος. Λοιπόν, να σας δώσουμε το λόγο στη, να δώσουμε το λόγο στη Σαμπίν. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν θέλατε να δώσουμε, να παρατείνουμε κάπως την προθεσμία πέρα από τις 4 του μηνός για την, ε, για την υποβολή τροπολογιών. Το συζητάμε μετά την παρουσία της Σαμπίνε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, διότι αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της ε, στρατηγικής, της ψηφιακής στρατηγικής της Ευρώπης και είμαστε επιτροπή που σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια και εξετάζουμε το θέμα. Ορίστε Σαμπίν. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόταση κανονισμού που μας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ο στόχο να έχει δώσει στον καταναλωτή πρόσβαση στο περιεχόμενο που έχει αγοράσει και στο εξωτερικό. Δηλαδή, ο καταναλωτής έχει αγοράσει την πρόσβαση σε μια υπηρεσία στη χώρα τους, έχει νόμιμη λοιπόν πρόσβαση σε αυτά, θα πρέπει να έχει και στο εξωτερικό πρόσβαση σε αυτό. Και το free to air το έχει αφαιρέσει από τη εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει όμως δυνατότητα καταχώρησης ή επαλήθευσης σε ό,τι αφορά το free to air τις υπηρεσίες αυτές. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν λοιπόν να συμπεριληφθούν και αυτές οι υπηρεσίες. Το περιεχόμενο θεωρείται στην περίπτωση αυτή ότι δεν εγκαταλείπει την έδρα του κράτους μέλους σε ό,τι αφορά αυτό τη διασυνοριακή πρόσβαση. Να μην ε, μπει από το παράθυρο, καταλαβαίνετε. Και έτσι να μην παραβιάζεται και η αρχή της εδαφικότητας. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή αρχή η οποία διαφάνεται σε, πολλές, σε πολλά σημεία της έκθεσης. Το θέμα λοιπόν της εδαφικότητας δεν το θίγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό το ότι τίθεται το θέμα αυτό από την Επιτροπή μας σε ό,τι αφορά θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, σου ταινίε, βίντεο κτλ. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι δομέ για την παραγωγή νέων περιεχομένων, η φορητότητα. Δεν σημαίνει α, διασυνοριακή προσβασιμότητα εδώ. Και αυτό το ξεκαθαρίζουμε σε μια τροπολογία την οποία υπέβαλα στο 12α, την αιτιολογική σκέψη, όπου υποδεικνύω με σαφήνεια ότι δεν μιλάμε για διασυνοριακή προσβασιμότητα μέσω ενός παραθυρακίου. Αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στην πολιτισμική ποικιλία που υπάρχει στην Ευρώπη ε, και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού αποτυπώνουν την ποικιλία και την πολυμορφία της Ευρώπης, δίνουν κίνητρα για τη δημιουργία νέων περιεχομένων και αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομευθεί από την οδηγία φορητότητας. Η φορητότητα λοιπόν έχει να κάνει με οπτικοακουστικά περιεχόμενα καταρχάς, Ισχύει βέβαια και για τη μουσική και για τα βιβλία και για τα πάντα, αλλά στην πράξη εδώ η διασυνοριακή προσβασιμότητα υπάρχει έτσι κι αλλιώς, γιατί για παράδειγμα τα βιβλία διατίθενται αναγλώσσα και στη μουσική υπάρχουν πανευρωπαϊκές άδειε πλέον και έτσι σε διάφορες περιπτώσεις υπάρχουν τέτοιες πανευρωπαϊκές άδειε και άρα δεν υπάρχει μεγάλη αλλαγή με την οδηγία αυτή, αλλά υπάρχει μεγάλη νομική βεβαιότητα αν ε, καταστούν φορητέ τέτοιε υπηρεσίε. Αυτό που είναι σημαντικό για τη λειτουργία της οδηγίας, θεωρώ, είναι ο σαφής ορισμός του κράτους μέλους ε, έδρας διαμονής. Εδώ βλέπετε είναι διαφορετικοί ορισμοί που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Και ήταν πάρα πολύ ασαφής ο ορισμός που περιλαμβανόταν στην πρόταση της οδηγίας. Στην έκθεση λοιπόν εισάγαγαμε έναν ορισμό που βασίζεται και σε νομολογία ε, του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του κ. Μαγδαλένα κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την οποία προκύπτει ότι σε τελική ανάλυση είναι ο ορισμός εκείνος κατά τον οποίο χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις ε, υπαλλήλου και για τις υπηρεσίες. Άρα θεωρώ ότι είναι σωστό να χρησιμοποιηθεί σε ό,τι αφορά το συνήθι τόπο διαμονής. Να είναι ο τόπος ε, όπου ε, βρίσκεται το επίκεντρο των δραστηριοτήτων, συναλλαγών του καταναλωτή και στο οποίο επανέρχεται τακτικά ο καταναλωτής και με τον οποίο έχει σύνδεσμο. Αυτό αφορά πολύ και τους ε, ανθρώπους που ταξιδεύουν, πολλοί που ζουν κοντά στα σύνορα, που κάθε μέρα τη σχέσουν τα σύνορα για να δουλέψουν σε μια άλλη χώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ε, το θέμα της φορητότητας να μην παρουσιαστεί ως πακέτο διακοπών μόνο. Όχι, είναι ε, ένα πολύ διαφορετικό πακέτο. Ο ορισμός λοιπόν του προσωρινού τόπου διαμονής αποτέλεσε αμφιλεγόμενο σημείο σε ό,τι αφορά τον ορισμό. Αυτό θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο. Γι' αυτό λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κάτι αντίστοιχο και αυτό αποτελεί το σημείο κλειδί της πρότασης προκειμένου να μην καλύπτονται μόνο ταξιδιώτε και αυτοί που πηγαίνουν διακοπέ, αλλά και οι φοιτητέ, αυτοί που δουλεύουν σε άλλο κράτο μέλο και πάρα πολλοί άλλοι από τη φορητότητα. Και επίσης ε, μας προβληματίζει και η ιδέα ε, του να αρχίσουν οι πάροχοι να μετράνε πόσε ώρε και πόσα λεπτά και πόσε ημέρε μένει κάποιο σε κάποιο άλλο κρατό μέλο και να αρχίσουν να μα παρακολουθούν. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει σαφή ορισμό ε, τη έδρα κατοικία. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το θέμα τη επαλήθευση ε, του κράτου μέλου κατοικία. Γιατί αυτό είναι σημείο κλειδί σε ό,τι αφορά την φορητότητα και συμφωνώ σε ό,τι αφορά τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το κράτος κατοικίας και τον έλεγχο, αλλά θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ελέγχονται τα συμφέροντά του και η τακτική ε, επιστροφή του. Όχι, θα πρέπει να γίνεται με άλλους τρόπους αυτή η επαλήθευση, με βάση τα κριτήρια αυτά, με βάση, συγγνώμη, τον ορισμό αυτό. Δεν θα πρέπει όμως ο πάροχος να αρχίσει να ελέγχει κατά πόσον και πώς ε, ζω στο σπίτι μου και πόσε ημέρε και μένω κτλ. Εδώ λοιπόν καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει παραδείγματα για τι δυνατότητε επαλήθευσή, Να αναπτύξει μια εργαλειοθήκη, ένα toolbox σο πράξεων και δεξιδότηση, προκειμένου να μπορεί να ενημερώνεται βάσει των τεχνικών εξελίξεων, χωρί να χρειάζεται διαρκώ να αναφέρουμε την οδηγία για την ε, φορητότητα. θα πρέπει να διασφαλίζεται νομικά ο δικαιούχος. σε περίπτωση που δεν γίνεται και σωστά από τον πάροχο η διαδικασία επαλήθευσης. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε στην οδηγία ο δικαιούχος σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται ε, σωστά ο έλεγχος του τόπου κατοικίας να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα αφαίρεση τη άδεια από τον παροχό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω σα είπα, θεωρώ ότι θα πρέπει να υποβάλει πιο συγκεκριμένα παραδείγματα για τι δυνατότητε επαλήθευση σε ένα προσάρτημα στα πλαίσια πράξεων καταξιοδότηση, προκειμένου να υπάρχει νομική βεβαιότητα για όλου του εμπλεκόμενου φορεί και για τον πάροχο τη υπηρεσία προκειμένου να ξέρει τι είδους μέθοδου, μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη σωστή επαλήθευση, για τον δικαιούχο, για τον πάροχο της ε, άδειας, προκειμένου να υπάρχει νομική σαφήνεια για το τι είναι μια σωστή μέθοδος ελέγχου και πού μπορούμε να παραπονηθούμε ότι δεν έλαβε σωστά δεν χώρα σωστή επαληθεύση και για τον καταναλωτή φυσικά από την άλλη πλευρά για να μπορούμε να του εξηγήσουμε με σαφήνεια ποια είναι η ένδρα κατοικία του. Και σε τι πλαίσιο μπορεί και επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες φορετότητα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, όπω σα είπα, καλό θα ήταν να αναπτυχθεί μέσω μιας εργαλειοθήκης, μέσω πράξεων κατά εξουσιοδότηση και με χαρά θα ήθελα να ακούσω και τις προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με παραδείγματα ενδεχομένω για τα νομικά κείμενα, να τα βάλουμε ίσω σε ένα προσάρτημα, σε ένα παράρτημα, να μπορούν αυτά να επεκταθούν ε, με πράξεις εξουσιοδότηση, για να μην ξανανοίγουμε συνέχεια το νομοθέτημα σε περίπτωση τεχνικών εξελίξεων. Για τις διευθύνσεις ε, IP. Θεωρώ ότι καταρχάς δεν είναι 100% αξιόπιστη ένδειξη για το έλεγχο τη ε, κατοικία γιατί υπάρχει και το VPN, η διευθύνση VPN. Και θεωρώ επίση ότι ούτε διαρκή και συνεχή έλεγχη θα πρέπει να υπάρχουν, γιατί αυτό θα σημαίνει διαρκή παρακολούθηση. Και θα ήθελα λοιπόν να μου υποβάλουν προτάσει εφόσον το επιθυμούν συνάδελφοι. Η προθεσμία ήταν 14η ε, Μαου. Αρχικά αυτό προβλεπόταν, αλλά μου φαίνεται πολύ σύντομο αυτό. Και γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλούσα να δώσουμε μία εβδομάδα παραπάνω προθεσμία. Μέχρι τις 11 Μαΐου διορθώνει η ομιλητρία. Γιατί είμαστε και πολύ... Είμαστε γενικώ στην Επιτροπή στην ώρα μας. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε. Καλό είναι να είναι καλοσχεδιασμένες οι τροπολογίε, να έχουμε το χρόνο μας με την ησυχία μας να αποβάλουμε τι προτάσει μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σαμπίν. Θα ακούσουμε και άλλου συναδέλφου όσον αφορά αυτή η πρόταση αναβολή Μπορούμε να αφήσουμε κάνα δύο μέρε. Αν αφήσουμε όμω 20 Ιουνίου την ημέρα που θα πρέπει να ψηφίσουμε ok anche io faccio la proposta di poter anche accogliere questa richiesta però lasciando naturalmente il voto in commissione Λοιπόν, 21 Ιουνίου θα ψηφίσουν την Επιτροπή και η Επιτροπή Γιούρι δεν έχει τοποθετηθεί βλέπετε ακόμα. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστές και στους σκιώδεις. Σκιώδεις και μετά συντονιστές. Όπως θέλετε. Ο κ. Γραμματικάκης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, όπως διαπιστώσατε και από τα όσα είπε η Σαμπίνα, θέλω να τη συγχαρώ, γιατί έκανε σπουδαία δουλειά και αυτό διευκολύνει και το δικό μου έργο. Πολύ το διευκολύνει. Η πρόταση βέβαια της Επιτροπής για τη διασφάλιση της διασυνορικής φορητότητας αποτελεί το πρώτο βήμα, αυτό είναι το δύσκολο, για τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Το κύριο είναι ότι αφορά, όπως και να το κοιτάξουμε, ένα μικρό σχετικά μέρος του πληθυσμού. Αν όμως γίνει μια ισορροπημένη και τεχνικά σωστή νομοθεσία, αυτό επιδιώκομαι, θα συμβάλλει ουσιαστικά, το τόνισε και η Σαμπίνα, στην επικείμενη αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, που έχει ασφαλώς πολύ μεγάλη σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο το γραφείο μου και εγώ πραγματοποιήσαμε μια σειρά συναντήσεων, κουραστικών συναντήσεων αλλά διαφωτιστικών με βασικούς φορείς που ενδιαφέρονται για το θέμα. Ενώ βέβαια συνεργαστήκαμε στενά με τους σοσιαλιστές συγητές από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών που έχουν ενδιαφέρον για τη φορητότητα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερο σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός θα αφορά τη φορητότητα ψηφιακών υπηρεσιών και όχι τη διασυνοριακή πρόσβαση, σε, ιδιαίτερα σε καλλιτεχνικό περιεχόμενο. Κάτι τέτοιο είναι φανερό ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιτεχνική δημιουργία και κυρίως, το τονίζω, στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Συνεπώς θέλω να στηρίξω πλήρως τις τροπολογίες της γήτριας υπαρθμό 2, 3, 4 και 5 που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Σκοπεύω μάλιστα αν διατηρήσω την ε, εγρήγορσή μου να καταθέσω και κάποιες επιπλέον προτροπολογίες που θα διευκρινίζουν νομίζω πλήρως το θέμα. Θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο σύμφωνα με την πρόταση του Συμβουλίου νομίζω ότι πρέπει να εισαχθεί ένα άρθρο που θα σπίζει την ξεκάθαρη υποχρέωση για τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν το κράτος μέλος διαμονής του συνδρομητή. Πιστεύω επίσης ότι μια ανοιχτή λίστα αποτελεσματικών μέσων επαλήθευσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην νομοθεσία. Η χρήση πολλαπλών μέσων μειώνει σημαντικά το περιθώριο κατάχρησης και συνεπώς προστατεύει τα δικαιώματα, αυτό θέλουμε όλοι, των δημιουργών σχετικά με το θέμα της προσωρινής παραμονής θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αναφερόμαστε σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το είπε και η συγκήτρια. Δεν πρέπει βέβαια να το καθορίζουμε επακριβώς για πολλούς λόγους αλλά και επειδή ο κάθε χρήστης έχει νομίζω διαφορετικές ανάγκες. Συμφωνώ τέλος με την πρόταση της συγγήτριας να αποσαφηνίσει τον ορισμό που αφορά το κράτος μέλος διαμονής Επίσης είναι φανερό ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα από έξι μήνες που πρότεινε η Επιτροπή για την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού. Κυρία Πρόεδρε, θα θυμηθώ το παλιό μου επάγγελμα που ήταν καθηγητής αστροφυσικής, όπως γνωρίζετε, και θα πω ότι αυτό το θέμα της φορητότητας ε, μου θυμίζει τον αριθμό των άστρων που βλέπουμε στον ουρανό με γυμνό μάτι, που είναι μόνο 3.000. Το θέμα όμως της όλης ψηφιακής πλατφόρμας είναι σαν επεκταθούμε σε ολόκληρο το γαλαξία που έχει κρατήσει την αναπνοή σας 200 δισεκατομμύρια άστρα, ίσως και παραπάνω. Αν μάθουμε όμως τον ουρανό μας καλά, θα διευκαλυθούμε και σε ολόκληρο το γαλαξία. Ευχαριστώ. Με αυτή τη λυρική έκφραση κλείνει η παρέμβαση. Και τώρα, συνάδελφε Σβέρ, ζητήσατε το λόγο, όχι. Λιούερ, έχετε το λόγο. Yeah, Ευχαριστώ. Ας ε, ε, πατήσω έτσι λίγο περισσότερο στη γη, αλλά νομίζω οι απόψεις μου είναι λίγο πολύ ίδιε με του προλαλήσαντες. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την έκθεσή της. Η ΣΥΑΡ τη στηρίζει και συχνά ε, συμφωνούμε και στηρίζουμε και ως ομάδα αλλά και ως ε, Βρετανική αντιπροσωπή στην ομάδα μας τέτοιου είδους προτάσεις. Το σημαντικό είναι να βρεθεί σωστή ισορροπία με έναν κανονισμό. Η φορητότητα επιγραμμικού περιεχομένου ως πρόταση πιστεύω κάποιο μουσικό ιντερλούδιο εδώ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα δώσει καταναλωτές ε, κάποια λογικά εύλογα δικαιώματα στην ενιαία αγορά, αλλά θα πρέπει οι πάροχοι υπηρεσιών να μην πέσουν θύμα υπερβολικών ρυθμίσεων και ο νέος κανονισμός να μην έρθει σε αντίθεση με τα εφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα, με την αρχή της εδαφικότητας ή την προστασία των δεδομένων. Και ιδίω ε, από την προοπτική της δικής μας Επιτροπής ε, Πολιτισμών, αυτός ο κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διατήρηση του δημιουργικού κύκλου, να μην υπονομευθεί ο κλάδος του περιεχομένου. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει ουσιαστικά ε, τη φορητότητα ε, να οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας ή της πρόσβασης. Θα θέλαμε λοιπόν ο κανονισμό να εφαρμόζεται ε, μόνο για όσου καταναλωτέ έχουν νόμιμη πρόσβαση σε περιεχόμενο που έχουν αγοράσει στη χώρα καταγωγή όταν βρίσκονται προσωρινά σε κάποιο άλλο κράτο μέλο. Επομένω, χρειάζονται οι σαφεί ορισμοί τόπο συνήθους διαμονή ε, και προσωρινή διαμονή για να υπάρχει και εμπιστοσύνη και προς τι επιχειρήσεις. Και θα πρέπει επίσης να δούμε κατά πόσο αν ε, αναφέρουμε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα αντιστοιχεί σε αυτή την προσωρινή διαμονή, αν αυτό λοιπόν θα βοηθούσε ή όχι τελικά. Νομίζω θα πρέπει να το, να το σκεφτούμε και να μην ε, βάλουμε αυτούς τους περιορισμούς τώρα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επαλήθευσης ώστε να έχουν κάτι των δικαιωμάτων ε, τη βεβαιότητα ότι μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν ε, καταβάλει τα ε, έχουν αγοράσει αυτό το περιεχόμενο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε μια άλλη χώρα. Θα πρέπει να δούμε πάλι τη χρησιμότητα αυτών των διαδικασιών, γιατί εξελίσσονται πολύ γρήγορα με την πρόοδο της τεχνολογίας, ε, άρα εξαρτάται πώς θα το δηλώσουμε στον κανονισμό, γιατί θα είναι δύσκολο ίσως να εφαρμοστεί ως κάτι νέο μετά. Και ξέρουμε με τις πηγές τεχνολογίας ότι είναι ε, κάποια πράγματα που γίνονται σήμερα που ούτε καν θα τα είχαμε σκεφτεί πριν από πέντε χρόνια και μάλλον το ίδιο θα συμβεί και στα επόμενα πέντε χρόνια, σε μια πεντετία από τώρα. Άρα εδώ λίγο θα διαφωνήσω με την άποψη κύριου Γραμματικάκη. Δεν θέλουμε επίση να υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο υπηρεσίε που παρέχουν ήδη φορητότητα, μουσική, παιχνίδια, ηλεκτρονικά βιβλία. Δεν λέω ότι δεν θα πρέπει να ε, μην ε, παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, ούτε πρέπει βέβαια και η πρόσβαση να μην είναι περιορισμένη. Αλλά πρέπει να τα προσέξουμε. Και το opt-in για τα free-to-air επίσης. Συμφωνώ με το σχόλιο του κυρίου Γραμματικάκη ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ό,τι αφορά τις περιόδους εφαρμογής για τις θεματεύσεις των συμβολέων. Δεν θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ περιοριστικοί. Ίσως είναι πολύ ε, μικρό το διάστημα των 6 μηνών. Δεν είμαστε αρκετά ρεαλιστικοί με αυτή την πρόταση. Γιατί δεν θα μπορέσουν να, γίνουν όσα πρέπει να γίνουν μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Επίσης, η ε, ελαστικότητα που θα πρέπει να προσφέρεται στους ε, παρόχους των υπηρεσιών. Έχουμε και κάποιες, ε, κάποιες άλλες παραμέτρους, σε αθλητικές οργανώσεις, Ολυμπιακοί αγώνες ή παγκόσμια πρωταθλήματα. Θα συνεργαστώ πάντως και με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για την σύνταξη μιας γνωμοδότησης που, αντίθετα με κάποιες άλλες πρόσφατες γνωμοδοτήσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι μια τάση αυτή τελευταία, ε, πιστεύω λοιπόν ότι με τη συνεισφορά όλων μας θα βελτιωθεί η έκθεση. Συνάδελφε Τόμ, Uh, thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Βαρχάιεν εμπεριέχει πολύ σημαντικές τροπολογίες και είναι καλή αρχή. Τονίζει το ότι η διασυνοριακή φορητότητα δεν είναι το ίδιο με την διασυνοριακή πρόσβαση. Η φορητότητα βασίζεται επί του νομικού ορισμού όπου ένας συνδρομητής θεωρείται ότι καταναλώνει από τη χώρα ε, του και όταν είναι στο εξωτερικό. Η δημιουργία αυτή, αυτού του νομικού σχήματος δεν επηρεάζει την εδαφικότητα των δικαιωμάτων. Στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως γίνονται παραπομπές στην ευρωπαϊκή πολιτισμική ποικιλομορφία. Όμως τα πλαίσια αυτό κάτι θα πρέπει να τονιστεί. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο online για μειονότητες. Οι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν περιεχόμενο το οποίο ταιριάζει στο γούστο της πλειοψηφία. Η μειονότητα από γειτονικέ χώρες Φερρυπίν πολύ συχνά δεν έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο της χώρας καταγωγής. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν νόμιμα, νόμιμες εναλλακτικές στις μειονότητες. Αυτό είναι εκτός του πεδίου εφαρμογή αυτού και δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικό, αλλά πρέπει να το επιστήσουμε, να επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα. Σαφέστερος ορισμός της χώρας διαμονής είναι κάτι που προτείνεται και είναι πρόσδεκτο. Σαφείς ορισμοί, όπως είπαν ήδη οι συνάδελφοι, θα μπορούσαν να αφορούν και τον όρο προσωρινό και τον πάροχο υπηρεσιών. Το προσωρινό είναι πέντε χρόνια, για κάποιους παρόχους υπηρεσιών είναι δύο εβδομάδες. Ένα επιχειρηματικό ταξίδι, Φερρυπίν. Ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ο ριζός του παρόχου υπηρεσιών online θα πρέπει να καθοριστεί σαφώς για να καθορίσουμε και τη φορητότητα. Πολλοί φορείς εμπλέκονται και θα πρέπει να εσαφίσω ότι πάροχη υπηρεσιών online είναι αυτό στον οποίο ο συνδρομητή έχει συνάψει σύμβαση με αυτόν. Προσωρινό μπορεί να θεωρηθεί ότι ορίζεται σαφώ για να αποφύγουμε τη διαφοροποίηση των χρονικών ορίων μεταξύ κρατών μελών. Τέλο. Λέγεται να, ότι πρέπει να δώσουμε κατ' εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιε πράξει για την εξακρίβωση μέσω εξοδότηση πράξεων μπορούμε τα μέσα επαληθεύσεως που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία δεδομένων εφαρμόζεται. Το σχέδιο γνωμοδοτήσεως προσθέτει σημαντικά πράγματα, χρειάζεται όμω δουλειά, ούτω ώστε τελικά στην πράξη να μπορεί να εφαρμόσουν τον κανονισμό. Αλλά συμφωνώ με του συναδέλφου που εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη προ την συγγήτρια για την έξοχη δουλειά που έκανε. Σα ευχαριστώ. Συνάδελφε Τρούπελ. Ναι, και από δική μου πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τη Σαμπίνε, γιατί όντω ε, είναι η καλή πρόταση αυτή που μα υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την διασυνοριακή προτεραιότητα. Και εγώ πιστεύω ότι σωστό είναι να το διακρίνουμε αυτό από τη γενικότερη διασυνοριακή πρόσβαση σε πολιτισμικά περιεχόμενα. Αλλά αυτό το έχει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και έθεσε ε, διαχωριστικέ γραμμέ. Όντω, ε, σε ό,τι αφορά το νομικό σκέλος, μπορεί κανείς ε, σε κάποιες περιπτώσεις ε, να πάρει μαζί το περιεχόμενο που έχει αγοράσει. Και αυτό δεν αγγίζει τα δικαιώματα του δημιουργού. Αυτό το έθιξε και στην προηγούμενη εβδομάδα σε μια ακρόαση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μια ομάδα ενδιαφερομένων, αλλά δεν συμφωνώ. Δεν είναι ότι έχουν πρόσβαση νέα άτομα, καινούργιοι άνθρωποι σε αυτό το περιεχόμενο. Όχι, απλά μπορώ να καταναλώσω το περιεχόμενο που έχω αγοράσει σε μια άλλη χώρα. Εγώ ω καταναλωτή ο ίδιο. Και Σαμπίνε, ε, έχεις δίκιο όταν λες ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει χρονικός περιορισμός σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην πληρωμένη συνδρομή, γιατί οποιαδήποτε τέτοιο περιορισμό θα οδηγούσε σε tracking, σε ελέγχους. Αυτό το απορρίπτουμε και εμείς ως λύση. Και θα ήθελα να τονίσω το εξή. Το θέμα τη χώρα ε, έδρα κατοικία είναι κεντρικό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει και ένα καθαρό ορισμό τη έδρα κατοικία και σαφή ορισμό ε, του πώ θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχο, η επαλήθευση. Είπες ε, καταρχά ότι έχει υπόψη να πράξει κατά εξουσιοδότηση, αλλά θα ήθελα να γίνεται και αναφορά στο νομικό κείμενο, στο διδακτικό του κειμένου. Είναι σημαντικό αυτό και πιστεύω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε κάποιε συγκεκριμένε προτάσει γιατί δεν θα ήθελα να τα αφήσω όλα να διευκρινιστούν μέσω πράξη κατά εξουσιοδότηση. Να προσθέσω επίση σε, σε ό,τι αφορά προσφορέ δημοσίου δικαίου, θα πρέπει να υπάρχει και μία λύση η οποία δεν θα είναι υποχρεωτική θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για κάποια μοντέλα συνδρομής, ένα opt-in ε, να υπάρχει δηλαδή ως μοντέλο, να μην προβλέπεται υποχρεωτικά, αν το επιθυμεί κανεί. Και τελευταία παρατηρήση παρά το γεγονό ότι το είπαμε ήδη και αυτά με τι ε, δυνατότητε επαλήθευση. και εδώ να μην προκύψουν μοντέλα tracking, παρακολούθηση, να βρεθούν άλλε λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν αφενός να συνεχίσει να αναπτύσσεται η ψηφιακή αγορά, να δίνονται ε, δυνατότητε στου καταναλωτέ, αλλά να μην περιορίζονται και τα ε, δικαιώματα του δημιουργού. Και να μην παραμένουμε όμω υπερβολικά και στην δυνατότητα ελευθερία, της ελευθερίας του καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σα ευχαριστώ. Συνάδελφε Κέστερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και σας ε, κύριε Συγκήτρια για την πρόταση αυτή και νομίζω ότι γενικά υπάρχει συμφωνία στην Επιτροπή μας ότι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορητότητα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να προωθηθεί η ενοποίηση της Ευρώπης ε, από οικονομικής απόψης είναι σκόπιμο και ωφέλιμο και ωφέλει και τους χρήστες και τους ε, δημιουργούς. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι είναι θετικό αυτό το βήμα, θετική αυτή η πρόταση και μπορεί να έχει και πολύ καλές ε, συνέπειες για όλη την Ευρώπη. Είναι σημαντικό να προσέξουμε ιδιαίτερα προκειμένου ο κανονισμός αυτός από πλευράς ε, του καταναλωτή να είναι διαχειρίσιμος, να μην είμαστε πάρα πολύ περιοριστικοί και πολύ αυστηροί. Και στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι κάνετε πολύ σκοπιμές προτάσεις ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη διάρκεια της παραμονής η οποία δεν θα πρέπει να περιορίζεται. Θεωρώ ότι αυτό είναι σκόπιμο και επίσης τονίζεται ότι δεν θα υπάρχει ε, παρακολούθηση των χρηστών. Νομίζω και αυτό πάρα πολύ σημαντικό είναι σε ό,τι αφορά το διάσταση της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας και των δεδομένων. Στο πλαίσιο μας αυτό έχω να κάνω μια ερώτηση. Εξηγήστε μας γιατί λέτε στην έκθεσή σας ότι θα ήταν απαραίτητο να γίνεται sampling, ε, δειγματοληψία των διευθύνσεων IP. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πώς θα γίνει στην πράξη. Ποιος θα κάνει αυτή τη δειγματοληψία. Ποιος θα κάνει τις έρευνες, ποιος θα πάρει τα στοιχεία, τα δεδομένα αυτά στη διάθεσή του και στη τελική ανάλυση ποιος θα πάρει την απόφαση. Τέτοιες ερωτήσεις λοιπόν ανακύπτουν σε ό,τι αφορά αυτό το sampling που αναφέρεται. Επίσης, πρότεινεται και διάφορα κριτήρια σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της έντρας κατοικίας. Για παράδειγμα, ε, τα τραπεζικά στοιχεία, τα φορολογικά στοιχεία, το φορολογικό αριθμό. Μήπως θα μπορούσαμε να τα περιορίσουμε όλα αυτά σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το δικαίωμα ψήφου. Αυτό έτσι εν είδη πρότασης. Λάβατε το υπόψη σας. Κάτι άλλο. Διατυπώνεται και κάποιες αμφιβολίες ότι δεν είναι δυνατόν ε, να έχει ο καθένας πρόσβαση στα φροντίδα αυτή μέσα σε ένα απλό σύστημα lock-in. Μα τι άλλη τεχνική λύση πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί. Θα πρέπει να το προβλέψουμε αυτό στον κανονισμό, θα δώσουμε ε, λευκή επιταγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αποφασίσει. Αυτές είναι οι ερωτήσεις ε, που ανέκυψαν κατά την ανάγνωση του κειμένου σας, το οποίο και θεωρώ καλό κατά τα άλλα. Ε, σας ευχαριστώ, η Πέτρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα είμαι σύντομη γιατί πολλά ακούσαμε ήδη από αυτά που ήθελα να πω. Νομίζω ότι όντω η οδηγία αυτή ήταν απαραίτητη ω πρόταση και κάνει καλή δουλειά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτά που πρότεινε η Σαμπίνα το στο κείμενό τη ε, συγκεκριμενοποιούν το κείμενο και χαίρομαι που δεν θα υπάρξει πιο στον ορισμό της προσωρινής διαμονής στο εξωτερικό ακριβώς λόγω του κινδύνου αυτού να υπάρχει δηλαδή ένας μόνιμος έλεγχος του χώρου διαμονής, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελεί το στόχο μας και το σκοπό μας. Ξέρω λοιπόν ότι σωστό είναι ότι δεν ε, ορίζεται πιο επακριβώς το ζήτημα αυτό. Αυτό που έχει να κάνει και που καθορίζει τα υπόλοιπα είναι ο τόπος κατοικίας. Γιατί δεν υπάρχουν και συστήματα αναφοράς σε όλα τα κρατη και θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει και ένα εύρος δυνατοτήτων επαλήθευσης ε, του τόπου διαμονής. Εγώ γενικά δεν είμαι υπέρ των πράξεων κατά εξουσιοδότηση, αλλά νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μια, ένα τεχνικό ζήτημα και μπορούμε να συμφωνήσουμε με πράξη κατά εξουσιοδότηση φυσικά υπό τον όρο ότι φυσικά θα τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανόνε για την προστασία των δεδομένων. Γιατί δεν μπορούμε αφενό να λέμε ότι δεν θέλουμε να ορίσουμε το χρονικό περιθώριο και από την άλλη να υπονομεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τον τόπο διαμονής. Σε ό,τι αφορά τον ε, αριθμό των τραπεζικού λογαριασμού, εδώ δεν είμαι πάρα πολύ διστακτική, γιατί όλοι όσοι έχουν κάποια πρόσβαση σε κάποιο φορητό περιεχόμενο έχουν δώσει μια πιστοτική κάρτα, ένα αριθμό λογαριασμού και αυτό περιλαμβάνεται στο προσωπικό του συμβόλαιο. Άρα εδώ πέρα δεν έχω πραγματικά αμφιβολίες. Αλλά ίσως καλό θα ήταν στο παράρτημα της οδηγίας να θέσουμε και να ορίσουμε κάποια από αυτά τα βασικά κριτήρια. Υπό ποιους όρους και πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια επαλήθευση του τόπου κατοικίας και μετά να τα αφήσουμε στην ευχαίρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να διτυπώσει δηλαδή τις λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω ότι ένα τέτοιο πλαίσιο καλό θα ήταν να τεθεί και στην οδηγία, αλλά όπως είπαν και οι συνάδελφοι, Όντω, να μην χρειάζεται να αναθεωρούμε την οδηγία κάθε φορά που θα ανακύπτει μια νέα τεχνολογική λύση. Δεν έχει νόημα. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή και σκόπιμη η προσέγγιση. Και σε ό,τι αφορά το free to air, τους δημόσιους και δυτικούς παρόχους, σωστά είναι αυτά που προβλέπονται και όντως ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ φορητότητας αφενός και μιας γενικής απογόρευση του γεωαποκλεισμού, αν το θέσω έτσι, αφετέρου. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στην οδηγία. Και έτσι λοιπόν υποστηρίζω τη σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Συνάδελφε Λιμπάτσικα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ την Σαμπίνα. Είναι έξοχη η έκθεσή της. Υπογραμμίζω κάτι που είπε η Σαμπίνα σε αυτή την Επιτροπή. Προωθούμε επανειλημμένα την κινητικότητα. Την κινητικότητα των νέων για τις σπουδέ, των νέων για να αποκτήσουν εμπειρίες, ε, να υποστούν ε, κατάρτιση. Το να παρέμβουμε για, την, για το μη περιορισμό της διάρκειας διαμονής. Με ανησυχεί αυτό που είπε ήδη η ε, Πέτρα. Ο κατάλογος που έχουμε παραμένει ανοιχτός των κατεξοδότησης πράξεων όσον αφορά τα μέσα εξακρίβωσης του τόπου διαμονής. Δεν είναι σίγουρα είναι ανοιχτός αυτός ο κατάλογος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και νέες δυνατότητες. Κατά την άποψή μου αυτή η λίστα θα πρέπει να καθοριστεί βάσει κάποιων θεμελιωδών παραμέτρων. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις. διευκρινήσεις θα ήθελα. Το πρώτο, κατανοώ απόλυτα το λόγο για το κείμενο που ανέφερε άνθρωπος Φεράιαν. Δηλαδή περνάμε από τον προσωρινό χαρακτήρα, τη χρονική διάσταση που είναι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής ε, ε, Επιτροπής, στο ξεπέρασμα το σιπίν του, του χρόνου που καθορίζεται με ένα ανώτατο όριο κλπ μέσω ενός καλύτερου ορισμού του τόπου διαμονής. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπε η συνάδελφος Πέτρα Καμερέβερτ, σε πολλές χώρες, όπως τη δική μου, μπορεί να πρέπει να ορίσεις πού μένεις και πού είναι η κατοικία σου, πού διαμένεις και πού είναι η κατοικία σου ίσως δεν καθορίζεται παρκώς ο τόπος δια, ε, διαμονής. Στην τροπολογία 12 λέει ότι τόπος όπου βρίσκεται το μόνιμο κέντρο συμφερόντων θεωρείται με χαρακτήρα διαρκή. Ίσως αυτό και ο τόπος συνηθισμένης διαμονής μαζί. Δύο όροι να πληρούνται δηλαδή. Έτσι να ερμηνευτεί. Διότι στο ιταλικό κείμενο Φαίνεται σαν να έχουμε δύο ξεχωριστά πράγματα. Και κάτι άλλο. Αν μπορεί να διευκρινίσει καλύτερα την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μπορεί να ξεπεράσουμε έτσι τον κίνδυνο να έχουμε μόνιμη διασυνοριακή πρόσβαση για τις κατεξουσοδότηση πράξεις. Προτιμάται αυτή η μέθοδος αντί να αναφέρεται στο άρθρο το θέμα των κριτηρίων που αναφέρονται ήδη στο κείμενο. Προσωρινά. Δεν είναι καλύτερο να καθορίζουμε κάποια κριτήρια γενικά, να είναι πιο γενική εφαρμογή και να είμαστε πιο σίγουροι τι έχει ο κανονισμός και να αφήσουμε στις κατεξουσοδότηση πράξεις καλύτερη προσαρμογή στις συνθήκες που δημιουργούνται να αφήσουμε τις γενικές συνθήκες στο κείμενο. Θα ακούσουμε μετά αυτά που είπα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα ακούσουμε τους συγητές. Η Μαρία Μαρτίν Πράτ έχει το λόγο, επικεφαλής της μονάδας DG Connect που έχει το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ την κυρία Φερχάιεν για μια εξαιρετική κατεμάς έκθεση. Επίσης, οι παρεμβάσεις των βουλευτών της Επιτροπής δείχνουν ότι είναι απόλυτα κατανοητή η στόχη που προσπαθεί να πετύχει με αυτή την πρόταση η Κομισιόν. Συμφωνούμε πλήρως με τα σημεία που επισημάνθηκαν ε, ως τα πλέον σημαντικά αρχίζει ενωμένης από την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ε, διαφορά μεταξύ φορητότητας και διασυνορικής πρόσβασης. Επίσης είναι σημαντικό να γίνει πιο σαφής ο ορισμός ε, του τόπου συνήθους διαμονής επίσης ότι δεν θέλουμε να περιορίσουμε την έννοια προσωρινή διαμονή το είπαν ορισμένοι βουλευτέ. Η πρόταση αυτή είναι σημαντική όχι μόνο για όσου είναι διακοπέ ε, σε κάποια άλλη χώρα, αλλά και για άλλου ανθρώπου. Βέβαια, έχουμε και την πρόκληση του πώς ε, θα εξασφαλίσουμε αυτή την επαλήθευση. Και έτσι έρχομαι και στα ζητήματα τα οποία εσείς ε, θέσατε με τις ερωτήσεις σας. Σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα την έννοια της συνήθως διαμονής Έχουμε την τροπολογία 12 του σχεδίου έκθεσης. Ε, λίγο πολύ αυτή είναι και η κατεύθυνση που ε, θέλουμε εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσουμε, δηλαδή να διευκρινίσουμε λίγο περισσότερο την έννοια αυτή και να την ορίσουμε, τη συνήθη διαμονή, όχι ως μια γενική έννοια, αλλά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, Διότι κάτι αντίθετο θα ήταν πολύ πιο πολύπλοκο και απαιτητικό, αλλά για τους σκοπούς αυτής, αυτού του κανονισμού να ορίσουμε τι θα πει συνηθής διαμονή. Και το δεύτερο, και έγιναν και κάποιες προτάσεις στην συγκητρία, επαλήθευση. Πώς θα ορίζεται επαρκώς και πώς θα επαληθεύει ο πάροχος τη συνήθη διαμονή. Είναι λίγο φαύλος κύκλος βέβαια το πώς θα γίνει αυτό και το πώς θα δοθεί επαρκής ε, σαφήνεια. Ε, μιλάμε για κανονισμό βέβαια. Άρα για όλα τα κράτη. Και τα κριτήρια θα πρέπει να είναι αξιόπιστα. Εμείς θέλουμε και κάναμε κάποιες προτάσεις ε, εκ των προτέρων. Δεν μιλήσαμε κατά της πράξη. Το Συμβούλιο μέχρι στιγμής στις συζητήσεις του δεν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο της πράξη. Απλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια ο κατάλογος των μέσων ε, επαλήθευσης να είναι ως το δυνατόν πληρέστερος και σαφέστερος. Και νομίζω ότι γι' αυτό θα απαιτηθούν ίσως και περαιτέρω συζητήσεις σε επίπεδο Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Το κατά πόσο τώρα εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει για μελλοντική επικαιροποίηση των μέσων επαλήθευσης ε, να έχουμε τη δυνατότητα κατεξοδότης πράξεων, θα πρέπει να δούμε και όχι μετά από ένα εξάμεινο, αλλά από την ίδια στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ αυτός ο κανονισμός, ότι οι υπάρχοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν αυτά τα μέσα παλήθευση. Ευχαριστώ, Ισαμπίν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, γενικότερη υποστήριξη στην προσέγγιση που επιλέξαμε για τις ερωτήσεις που κάνατε και θα ήθελα να αναφέρω και να απαντήσω σε κάποια σημεία. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το θέμα της δειγματοληψίας των διευθύνσεων IP, αυτό είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια δυνατότητα και για τις ε, συμβάσεις που υπάρχουν με άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα με τηλεφωνικές υπηρεσίες. Αυτό ήταν στο εντελογική σκέψη 17 έως τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το αφαίρεσα από την εντελογική σκέψη γιατί ήθελα πιο σωστή και καθαρή, καθαρό ορισμό για την επαλήθευση μέσω εργαλειοθήκης. Ε, φυσικά αυτή η εργαλειοθήκη μπορούμε να θα συμφωνήσουμε κατά πόσον θα τη γνωρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω πράξη κατά Αυτό που με απασχολεί είναι να υπάρχει νομική βεβαιότητα για όλου του εμπλεκόμενου φορεί. Προκειμένου να υπάρχει ένας σωστό και καθαρός ορισμός σε ό,τι αφορά τον τόπο κατοικία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μόνο μία μέθοδο και να συμπεριληφθεί μόνο μία μέθοδος, γιατί, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ε, μήτρο πρώτης κατοικία σε κάθε κράτος μέλος. Ε, για παράδειγμα, εγώ μπορεί να έχω πολλά σπίτια και πολλούς, ε, πολλούς αριθμούς τηλεφώνου. Πού είναι η πρώτη μου κατοικία. Γι' αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να μην υπάρχει αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, να υπάρχει σαφής ορισμός. Και να πω ότι στο σημείο αυτό ειλικρινά δεν μπορώ να ορίσω την δυνατότητα επαλήθευση για 28 κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να υπάρχει αυτή η ελευθερία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν για παράδειγμα ένα κράτος ε, ιδρύσει μήτρο τέτοιων κατοικίας, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Να υπάρχει ένας ξεκάθαρος τρόπο. να βρεθεί δηλαδή ε, θα ήταν καλό να βρεθεί βέβαια και μια μέθοδο επαλήτευση η οποία τεχνολογικά να επιτρέπει σε όλου να τα χρησιμοποιήσουν, αλλά ε, να συνεργαστούμε στο τομέα αυτό. Να το βάλουμε ενδεχομένω ε, στο παράδειγμα, δεν έχω αντίρρηση, αλλά να μπορεί να επεκταθεί στη συνέχεια. Να μην είναι χρειαστεί να ανοίγουμε κάθε φορά την οδηγία σε περίπτωση που, για παράδειγμα, θέλουμε να προσταθούν κάποια εργαλεία στην εργαλειοθήκη ε, στο παράδειγμα. Να μπορεί μέσω πράξης κατά εξουσιοδότηση να επεκταθεί αυτή η εργαλειοθήκη. Νομική σαφήνεια πάντα πρέπει να υπάρχει. Σε ό,τι αφορά τις παροχές free to air. Καλό είναι να υπάρχει αυτή η σύνδεση με τον πελάτη και γι' αυτό λοιπόν ζήτησα το τέλος, ε, το ραδιοφωνικό τέλος, το οποίο δεν συνδέεται απαραίτητα α, με, τα, με τις ραδιοφωνικές εκπομπές, να μην έχει τέτοια σχέση για να υπάρχει τέτοια σαφήνεια σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτές τις ελεύθερες πρόσβασης υπηρεσίες, τις free to air. σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την κρυπτογραφημένη αποστολή ε, περιεχομένου, γιατί υπάρχουν κάποια κρατημέρια που το κάνουν αυτό, θεωρώ ότι εκεί πέρα υπάρχει μια άμεση σχέση, γιατί έχουμε τη διεύθυνση αυτή. Και αυτό είναι μια ευκαιρία, όχι υποχρέωση. Αν ε, υπάρχει αυτή η επαλήθευση μια τέτοια εργαλειοθήκη, ε, θεωρούμε ότι πληρούμε όλα αυτά τα κριτήρια. Γιατί να μην υπάρχει λοιπόν, λοιπόν δυνατότητα φορητότητα. Άρα να συμπεριληφθούν αυτές οι υπηρεσίες. Γιατί όχι, γιατί δεν συνεπάγονται επιπλέον έξοδα και τέλη. Ούτε αγγίζουν ε, τα θέματα αδειών. Γιατί ουσιαστικά καλύπτουν την ίδια επικράτεια που κάλυπταν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει δηλαδή επέκταση, αλλά ουσιαστικά καλύτερα αξιοποιήσει αυτό που αποκτήθηκε νόμιμα. Όπως σας είπα, χαίρομαι στο σημείο αυτό. Γιατί ελπίζω ότι θα καταλήξουμε στη συμφωνία σύντομα σε ό,τι αυτά τα σημαντικά στοιχεία. Όπως σας είπα, σημαντικό να μην υπάρχει χρονικό περιθώριο. Δεν μπορούμε να ορίσουμε, θεωρώ, πόσες ημέρες, πόσα χρόνια. Α, τότε το σημείο, δηλαδή, στα πέντε που έχω μετακομίσει σε μια άλλη χώρα που θα πρέπει να θεωρείς ότι έχω αλλάξει τόπος κατοικίας. Αυτό είναι σαφές, αλλά όταν πάω για έξι μήνες ε, στην Ισπανία για να κάνω εράσμους, ουσιαστικά η πρόσβαση, η πρόθεσή μου είναι να επιστρέψω. Ε, αν τώρα συναντήσω το μεγάλο έρωτα ή αποφασίσω και βρω μια δουλειά να μείνω στην Ισπανία, εντάξει, θα αλλάξω και το τόπο κατοικίας μου. Αλλά νομίζω ότι τέτοιες λεπτομέρειες θα πρέπει να τις έχουμε συνοηθεί. Και σε ό,τι αφορά το σαφή και ξεκάθαρο ορισμό του τόπου κατοικίας. Γι' αυτό ακριβώς βάσισα τον ορισμό αυτό σε απόφαση του δικαστηρίου για τους Ευρωπαίους ε, υπαλλήλους. Γιατί αυτό ήταν το θέμα που πραγματεύτηκε η νομολογία. Τι είναι Ποιο είναι ο τόπο κατοικία, οι πέντε μέρε που δουλεύω στι Βρυξέλλε ή όταν θα πηγαίνω για παράδειγμα στην ε, χώρα μου να ζήσω το Σαββατοκυριακό. Και τι γίνεται για παράδειγμα όταν μετακομίσει και η οικογένειά μου. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειε οι οποίε θα πρέπει να οριστούν ξεκάθαρα. Για να υπάρχει βεβαιότητα. Και το τονίζω, όχι για το σκοπό του να ελέγχει και να υποχρεούνται να ελέγχει ο πάροχος της υπηρεσίας όλα αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά να υπάρχουν σαφείς ορισμοί σε περίπτωση νομικής διαφωνίας. Και θεωρώ ότι εδώ μπορούμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις στις οποίες θα δεχτεί και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων προκειμένου να ακουστεί μια ομόφωνη φωνή από πλευρά του Κοινοβουλίου και προβλέπω στην καλή συνεργασία με τους Κιώδες και τους υπόλοιπους συναδελφούς. Ευχαριστώ. Ναι, Ευχαριστώ Σαμπίνε. Λοιπόν, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, αν συμφωνούμε, είναι 11 Μαΐου στις 11, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της του συνάδελφου Γιάννη Γκάιερ, μάλλον, που είναι εισηγητή για τον προπολογισμό του 2017, ο κύριος Γκάιερ. Του ευχόμεθα καλή τύχη για αυτή την προσπάθεια. Περνάμε σημαντική ε, περίοδο για το διάμεσο του προγραμματισμού και στα πλαίσια των συναντήσεων που έχει ο κ. Γκάιερ με όλες τις επιτροπές. Τον ευχαριστούμε που ήρθε και εδώ να συναντηθεί με την Επιτροπή Πολιτισμού για να συζητήσουμε τις πρωτοβουλίες του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Η Επιτροπή, όπως γνωρίζετε, θα παρουσιάσει τον το σχέδιο προϋπολογισμού τέλος Μαΐου. Λοιπόν, αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης με αυτή την συνάντηση είναι κάτι που δρομολογεί της Επιτροπή όσον αφορά τον προπολογισμό του 2017. Θα δώσω απαραίτητη το λόγο στον κύριο Γκάιερ. Ζητώ συγγνώμη, τον κάναμε περιμένει κάποια λεπτά. Και μετά ε, στους συγγητές, τον κύριο Στρογεύσκη και τους και συγγητές και σε όλους τους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν για το θέμα. Ένα δεκάλεπτο θα έλεγα, έχετε το λόγο. Αν χρειαστείτε λίγο παραπάνω, δεν ξέρω. Με τα χαράς να ακούσουμε την παρουσίασή σας λοιπόν. Ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστώ για, φιλική, για το φιλικό χειροτερισμό. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, όντως διατρέχω όλες τις επιτροπές ως ε, εισηγητής ε, για το Γενικό Προϋπολογισμό του 2017 για να μαζέψω τις εντυπώσεις των επιτροπών και αυτή η προσεκτική διατύπωση νομίζω ότι προδιαθέτει και προϋποθέτει ότι δεν θα μπορέσω ενδεχομένω να ικανοποιήσω όλα τα δεκτήμα σας. Αλλά θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω την ε, τοποθετησή μου σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Το η κυρία Πρόεδρος αναμένουμε το σχέδιο του προϋπολογισμού στις 25 Μαΐου. Όσο δεν έχουμε στη διάθεσή μας την πρόταση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, συζητάμε λίγο στον αέρα. Μπορούμε να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε για τον προϋπολογισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ποια θα είναι τα γενικότερα πλαίσια. Σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 6 εβδομάδες στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο έδωσε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και εκεί λοιπόν αναφερόταν το τι περιμένουμε από τον προπολογισμό αυτό. Αυτό ως γενικότερη κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά ασφαλώς πρόκειται και για ένα έγγραφο το οποίο δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένο γιατί το αντικείμενο της αντιπαράθεσης δεν υπάρχει ακόμα. Δεν το έχουμε ε, Και το Συμβούλιο δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές και οι συνάδελφοι από το Συμβούλιο έκανε την κατάσταση λίγο πιο απλή. Έξι σελίδες ε, περιλαμβάνει το έγγραφο και ουσιαστικά μια μισή πρόταση είναι καινούργια. Τα υπόλοιπα είναι κοπιπέστα από προηγούμενη χρονιά. Τώρα βέβαια δεν έχουν και άδικο απόλυτα. Συμβούλιο ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και εδώ είναι το πρώτο σημείο το οποίο θα ήθελα να θέξω σε ό,τι αφορά και τη σημερινή μας συζήτηση. Φυσικά, όλες οι κρίσεις ε, που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε στο σχέδιο προϋπολογισμού για το τρέχον έτος, το 2016, όλες αυτές οι κρίσεις λοιπόν συνεχίζονται δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί θα υπήρχε οποιοδήποτε λόγος. Τα, τις υψηλές δαπάνες τις οποίες ε, εγκρίναμε, κινητοποιήσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για ποιον λόγο λοιπόν ε, οι δαπάνες αυτές για την ε, υποστήριξη της αντιμετώπισης της κρίσης, γιατί θα έπρεπε να περιοριστούν οι δαπάνες αυτές ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός προβλέπει πάνω από 5 δις στις κατηγορίες 3 σε ό,τι αφορά ε, την πολιτική και στην κατηγορία 4, την εξωτερική πολιτική, για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης με τον ένα τρόπο ή για την καταπολέμηση ε, των, ε, της ρίζας ε, της ε, μετανάστευσης, ό,τι αφορά λοιπόν την κατάσταση των προσφύγων στις ε, γειτονικέ χώρες, στη Συρία, στο Λίβανο, στην Τουρκία, στην Ιρλανδία. Και νομίζω αγαπητοί συνάδελφοι όλοι βλέπουμε ειδήσει. Ε, κανείς ε, εδώ πέρα δεν φαντάζομαι να έχει στηρίξει όλους τους τις ελπίδες στην διαδικασία στη Γενέβη. Ελπίζουμε να υπάρχει κάποια δυνατότητα κατάπαυση πυρός στη Συρία και μια μελλοντική διάσταση ειρηνευτική διαδικασία, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι η κρίση αυτή θα τερματιστεί σύντομα και μαζί τη και η προσφυγική κρίση. Άρα δεν βλέπω να υπάρχει κανένα λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του 2017 για τι κατηγορίε αυτέ 3 και 4. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό στον προπολογισμό και αυτό γιατί συμπεριλαμβάνεται και από την κατηγορία 3 για την αστρική πολιτική ένα κομμάτι. Και ένα κομμάτι δεν διατίθεται σε ό,τι αφορά την ε, καταπολέμηση της κρίσης της προσφυγικής. Για να ενισχύσουμε αυτά που θα θέλαμε να ενισχύσουμε και σημαντικά προγράμματα τα οποία έχουμε, στα οποία έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Αυτές είναι οι συνθήκε πλαίσιο. Η οικονομική κρίση, την οποία έχουμε συζητήσει σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εξέλθει αυτή τη οικονομική κρίση με ικανοποιητικό τρόπο. Φυσικά τα πράγματα διαφέρουν ανά χώρα σε χώρα, αλλά συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι και λαμπρή η κατάσταση σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση. Ό,τι έχουμε καταβάλει λοιπόν ω προσπάθεια από πλευρά του προπολογισμού για τη βελτίωση τη ε, της κατάστασης και όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν δεν μπορούμε να τα μειώσουμε. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. 8 ευρώ έχουμε, θα πρέπει να βάλουμε στην άκρη στον προϋπολογισμό για να έχουμε ε, την εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Ταμείο, το ΕΦΣΥ. Τα χρήματα αυτά δεν έχουν συμπληρωθεί στις γραμμές του προϋπολογισμού και εδώ λοιπόν έχουμε για τα οποία ρέουν προς μία πλευρά την οποία θα πρέπει ασφαλώς να λάβουμε υπόψη. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν, τουλάχιστον θεωρώ εγώ, ότι το μεσοπρόθεσμο χρηματοοικονομικό πλαίσιο στα κρατημέλη για τα έτη 2014 και εξή ήταν ε, κενά λόγια. Με το μεσοπρόθεσμο λοιπόν αυτό το πλαίσιο καταρχάς μειώθηκε η σύμβολη των κρατών μελών 1% ήταν το ποσοστό αυτό ανάλογα με το ΑΕΠ και αυτό ε, χαροποίησε πολλά κράτη-μέλη και ιδιαίτερα την ε, Γερμανία. Αλλά διαπιστώνουμε ότι τα χρήματα πολύ απλά δεν φτάνουν. Το 2014, 2015 2016 είναι η τρίτη, ο τρίτος προπολογισμό που καταρτίζουμε στο πλαίσιο αυτού του δημοσιονομικού πλαισίου και πολύ απλά δεν φτάνουν τα χρήματα που διαθέτουν τα κράτη-μέλη. Στα τέλη του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης. Το Κοινοβούλιο πάντα επέμενε για την αναθεώρηση. Δηλαδή τα ελέγχουμε όλα, τα βάζουμε κάτω και βλέπουμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί. Τα κράτη-μέλη λοιπόν μιλούσαν πάντα μόνο για μία αναθεώρηση. Και επιμένουν σε αυτό, δηλαδή να κάτσουμε, να κοιτάξουμε κατά πόσο λειτουργούν τα πράγματα και κατά πόσο δεν λειτουργούν και αν δεν λειτουργούν, εντάξει, να εξαγάγουμε συμπεράσματα, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο 2020 και μετά. Στην πολιτική λοιπόν αυτή η κατάσταση και στο πολιτικό αυτό πλαίσιο θα διεξαχθούν οι συζητήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσει να αναπτύσσει τη θέση του ε, για την αναθεώρηση και θα πρέπει φυσικά αυτό, αν συμβεί αυτό, θα υπονομεύσει και τι συζητήσει για τον προπολογισμό. τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε στον προϋπολογισμό θα πρέπει να συνδέονται πιο πολύ ε, με τα οικονομικά έγγραφα της, της Ευρώπης. Έχουμε ε, ετήσια έκθεση ανάπτυξης, για παράδειγμα, ευρωπαϊκή οικονομική προοπτική. Μιλάμε στο εξάμεινο για τις δυνατότητες προσαρμογής των κρατών μελών. Και όντως θα ήταν απτή η ευρωπαϊκή υπεραξία αν συνδέαμε τα έγγραφα, τα εργαλεία αυτά με τις οικονομικές αυτές προβλέψεις. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Νεολαία, για την απασχόληση της νεολαίας θέλουμε να συνεχιστεί και αποφασίσαμε να υπάρχουν κάποιες θέσεις μαθητείας. Δεν μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε επιπλέον πόρος και τα κάτι μελη επί της αρχής. Πώς να το διατυπώσω προσεκτικά, επί της αρχής δήλωσαν ότι ήταν πρόθυμα να συνεχίσουν σε ό,τι αφορά αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Νεολαία, αλλά θέλουν καταρχάς να γίνει αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει ακόμα αυτή η αξιολόγηση, δεν τίθεται. Αν είναι θετική η αξιολόγηση αυτή, αν αυτό δηλαδή αποδείξει ότι στις χώρες αυτές όπου η κατάσταση είναι δραματική, υπάρχει απτή βελτίωση της κατάστασης για τους νέους ε, θέλουν να συνεχίσουν. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Εμάς ε, στο Κοινοβούλιο μας απασχολεί η καταπολέμηση της ένδυας. Ε, δεν είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στις κατευθυντήριες γραμμές νομίζω ότι έχουμε θέσει προτεραιότητα, ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της φτώχειας μεταξύ των παιδιών και θα πρέπει στις συζητήσεις στα εκάστοτε κρατή-μέλη να λεφτούν υπόψη και οι ειδικέ συνθήκες. Και εδώ θα περάσω στο πολιτικό σκέλο. Αν το Κοινοβούλιο αφενό ε, θέλει να, υπάρχουν, να υπάρχει ενοποίηση του προπολογισμού, αλλά μια διαφορετική προτεραιότητα ε, με ε, πλειοψηφία θέλει να κάνουμε πιο πολλά με τον ίδιο ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούμε δηλαδή να ζητάμε τα κρατημέλη να μην ξοδεύουν χρήματα και να κάνουν έτσι, οικονομίες και από την άλλη να τους ζητάμε πιο πολλά χρήματα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Θα πρέπει να δούμε πού βρίσκονται οι πολιτικές προτεραιότητες. Όντως υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας. Δεν λέω. Το θέμα όμως που έθιξα πέρασε, και μάλλον δεν πέρασε με πολύ ωριακή πλειοψηφία σε ό,τι αφορά τι κατευθυντήριε γραμμέ. Και πρέπει να αποφασίσουμε, εν πάση περιπτώσει, τι θέλουμε, να τοποθετηθούμε. Η κατάσταση σε ό,τι αφορά τι πληρωμέ έχει κάπω χαλαρώσει. Έχουμε απλήρωτους λογαριασμούς, τώρα πλέον έχουμε νέο χρήμα στον προπολογισμό και έτσι μειώνεται ο αριθμός των απλήρωτων λογαριασμών. Είναι πολύ τεχνική τη δικασία αυτή, δεν θα σας ε, κουράσω. Η πρόβλεψή μου και η πρόβλεψη όλων των οικονομολόγων ε, είναι ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο γιο-γιο, δηλαδή μειώνεται τώρα, θα αυξηθεί μετά πάλι το ποσό αυτό. Χρησιμοποιούμε χρήματα για να πληρώσουμε λογαριασμού, αλλά όταν ε, φτάσουμε στο τέλος της χρηματοοικονομικής περίοδου θα μας ε, τελειώσουν τα λεφτά. Προς το 2020 δηλαδή και πάλι θα έχουμε έτσι μεγάλο κύμα απλήρωτων λογαριασμών. Αυτό δεν ε, σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, απλά ήθελα να σας το αναφέρω σε κάθε περίπτωση. Στους συντονιστές στην Επιτροπή Προπολογισμού, στην οποία θα πρέπει να επιστρέψω άμεσα, το συζητήσαμε το θέμα, αυτό, το θέμα αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει έναν προπολογισμό που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα. Focused on results. Αυτό δεν θα παίξει κάποιο ρόλο για τον τρέχοντα προπολογισμό, γιατί τα πιο πολλά προγράμματα που έχουμε αποφασίσει από ό,τι ξέρετε είναι πολίτη και φυσικά δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε κάτι ε, σε ένα έτος, ούτε να προσμετρήσουμε τα αποτελέσματα ενός πολιτικού προγράμματος, αλλά αυτό το, αυτή η εστίαση στα αποτελέσματα θα αποτελέσει κριτήριο για τα προγράμματα του Συμβουλίου. Για το Εράσμος, ε, για παράδειγμα, Ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ασφαλώς, γιατί ε, όλα είναι εξαιρετικά. Η εφαρμογή και τέτοια προγράμματα χρειάζομαστε. Και κλείνοντας να πω ότι εγώ θεωρώ ότι το πρόγραμμα Erasmus ε, έχει μια ευρωπαϊκή υπεραξία η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί. Είναι προφανέστατη. Τώρα αυτό κατά πόσο θα ισχύει για κάθε περιφερειακό και λοιπό πρόγραμμα, εδώ μπαίνει ερωτηματικό. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει και κάθε επιτροπή. Αλλά θεωρώ ότι ήταν και ενδιαφέρον να το κάνει αυτό η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Αλλά από άποψη αποτελέσματος ε, θεωρώ ότι είναι ξεκαθαρά τα πράγματα και εγώ σε κάθε περίπτωση σα υποστηρίζω. Ευχαριστώ πολύ. σα ευχαριστώ για το ειλικρινές και άμεσο ύφο σα ε, και τι διάφορε πολιτικέ πτυχέ που αναφέρατε. Πάντα αντιμετωπίζουμε δυσκολία να αντιμετωπίσουμε ανοιχτά το περιορισμό που επιβάλλει ένας προϋπολογισμός που περνά περίοδο μεγάλων κρίσεων και πετούνται νέοι πόροι λόγω νέων πολιτικών και πρέπει πάντα να παίζουμε τους ίδιους πόρους, μειώνοντας ίσως τους πόρους άλλων προγραμμάτων. Αυτό συνέβη στα δικά μας προγράμματα, το θέσαμε όπως ε, γνωρίζετε και στο Εράσμος και στη Δημιουργική Ευρώπη η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την κρίση των προσφύγων την κρίση της ζωσβαστικοποίησης, της απαιτήσει για την ένταξη, την εκπαιδευτική και τη μεγάλη πολιτισμική πρόκληση που υπάρχει, ε, λάβαμε υπόψη ότι ίσως στις 10 προτεραιότητες η λέξη παιδεία και πολιτισμός απουσιάζουν και θα πρέπει να αποκληθούν σήμερα η ανδέκατη προτεραιότητα. Αυτό πιστεύουν και αρκετά κράτη-μέλη. Αντίθετα, βλέπουμε ότι όσον αφορά τις νέες απαιτήσει, οι οποίες είναι σημαντικότατες, ε, περικόπτονται τα χρήματα από προγράμματα που ήδη υφίστανται. Θα πρέπει μαζί να πολεμήσουμε και αυτό. Και σαφώς το θέμα ουσιαστικά πολιτικό είναι του προπολογισμού της ενώσεως που εξακολουθούμε να βάλουμε από χρόνο σε χρόνο. Και βλέπουμε ότι αυτό δεν επιτρέπει να αναπτύξουμε ευρωπαϊκές πολιτικές, πλήρως ευρωπαϊκές. Θα δώσω το λόγο, ευχαριστώντας σας για την εισαγωγή, σε τέσσερις συναδέλφους που ζήσαν το λόγο, δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλοι. Ξεκινώ. Α, συνάδελφος Ροζιέσκη έχει καθυστερήσει, δεν ξέρω αν θα προλάβει να μείνει για λόγους ε, της... Με τους Κιώδης θα ξεκινήσουμε. Συνάδελφε Σβέρ, Τρούπελ, Μόργανο και Λιούερ έχουν ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Γιένς Γκάιερ. Ήταν έξοχη η παρουσίαση που έκανε όσον αφορά τα δημοσιονομικά ζητήματα Έχουμε συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά το Erasmus Συν. Είμαι συγητή για το Erasmus Plus και θα ήθελα με ενδιαφέρον να έχω σαφή στοιχεία όσο πιο επακριβή γίνεται. Η αναθεώρηση αναφέρθηκε του προϋπολογισμού για φέτος. Επ' αυτής της ο προϋπολογισμός του 2017 θα καταρτιστεί. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να γνωρίζω ποια θα είναι η αύξηση ε, ποια θα είναι η αύξηση του χρόνου στον αφορά το Erasmus ε, Συν για τον επόμενο χρόνο. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Helga Truppel. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Γιάννη Σκάιερ για την παρουσίαση αυτή που μα έκανε. Την παρουσίαση όλων αυτών των προκλήσεων, των προβλημάτων που έχουμε σε ό,τι αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Όταν αποφασίσαμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, κάτσαμε και συζητήσαμε από τότε ότι ήταν πολύ περιορισμένο. Για πρώτη φορά μειώθηκε στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σαφέ ε, για όλου το Κοινοβούλιο. Ακόμα και αν συμφωνήσαμε τελικά σε αυτό το κακό σημείωμα ότι ήταν κάτι το οποίο επικρίναμε, γιατί είχαμε πει ότι θα καταλήξουμε τελικά μοιραία σε μια κατάσταση που πολύ απλά δεν θα φτάνουν τα χρήματα για τα προγράμματα όλα. Επίσης επικρίναμε το ότι συνέχιζε να μην υπάρχει επαρκή ευελιξία στον πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό ακόμα μας βασανίζει. Να κοιτάξουμε τα μεγάλα προγράμματα, το Erasmus ε, Plus. Το είπε, ε, το είπε και εσύ, Γιάννης ε, Ήταν πάρα πολύ επιτυχία το πρόγραμμα αυτό και πραγματικά δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος να μην το επεκτείνουμε το πρόγραμμα αυτό. Ο αριθμός των φοιτητών, των νέων επιχειρήσεων, των ατόμων που επωφελούνται και μαθαίνουν για μια ολόκληρη ζωή. Αυτό λοιπόν ε, μα οδηγεί στο ότι θα έπρεπε να αυξηθεί ο προπολογισμό. Το ίδιο και για το Creative Europe. Ξέρουμε ότι είναι ένα αρκετά μικρό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και όλοι, όλα τα στοιχεία μας οδηγούν στο ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πολιτισμική ανταλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Πολίτη μειώθηκε μάλιστα σε ό,τι αφορά το πολίτες πλαίσιο. Είναι πραγματικά αντιπαραγωγικό και αντίθετο αυτό με τους στόχους που έχουμε θέσει για το ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να έχουν σε επαφέ πέρα από τα σύνορα οι πολίτες να χτίζουν καινούργια προγράμματα κτλ. Αντίθετα λοιπόν με αυτά που ήθελε να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ε, επαφή μεταξύ των πολιτών. Κάτι άλλο που ήθελα να δείξω σε ό,τι αφορά την υποβολή αιτήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις ακούμε ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκη η διαδικασία υποβολη αίτηση και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά μικρά ποσά. Είναι δυσανάλογο ο αριθμο των εγγράφων που πρέπει να συμπληρωθούν. Θα ήθελα λοιπόν να σα παρακαλέσω να το θέσουμε αυτό το θέμα όταν θα κάνουμε τη διαπραγματεύση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην αποτρέπεται τελικά ο κόσμο και να αποθαρρύνεται, ιδιαίτερα για τα μικρά αυτά έργα τα οποία θέλουμε να προαχθούν. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει. Τελευταίο σημείο. Θα πρέπει τα προγράμματά μα να τα αξιολογήσουμε για τους πολίτες και να τα χρησιμοποιήσουμε και για τους πρόσφυγες και για την αλλαγή μεταξύ των πολιτών. Και αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ίσως στο τέλος θα πω κάτι, συνάδελφε Μοργάνο. Ευχαριστώ ιδιαίτερος τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Είμαι στο μήκο κύματο αντιπροέδρου της κυρίας Τρούπελ. Όσον αφορά κάποια θέματα που υπογράμμισα να τονίσω και εγώ. Έχουμε πολλές κρίσεις Χρειάζεται συνέχεια επενδύσει στον τομέα της παιδείας, επαγγελματική καταρτήσεω και νεολαία. Αυτό διότι μέσω αυτών των προσπαθειών σήμερα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Όταν στα πλαίσια του προπολογισμού, όσον αφορά την Επιτροπή Πολιτισμού, ε, δίνονται λιγότερα. Ε, υπάρχει αντίφαση. Στα κοινοβουλευτικά κείμενα τελικά μειώνονται, ζητούνται μειώσεις των πόρων. Πολλά προβλήματα πλήττουν την Ευρώπη του τελευταίου μήνε. Μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα μόνο αν έχουμε αποφασιστικότητα για μια πιο πανευρωπαϊκή προσέγγιση που ακολουθεί και τον πειραματισμό και την καινοτομία σαν κατεύθυνση. Σημειώνονται η συμπληρωματικότητα και η συνεργασία μεταξύ φεσταμένων προγραμμάτων με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή μα. Κυρίω τα έχουμε το Erasmus Plus, τη Δημιουργική Ευρώπη, η Ευρώπη για του πολίτε, και έχουν τεθεί προτεραιότητες ε, κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Ανάπτυξη επενδύσεις όπως ε, υπενθυμίστηκε και σωστά από τον εισηγητή. Ανάπτυξη και επενδύσεις για να αντιταχθούμε στην ανεργία, κυρίως στην ανεργία των ε, νέων. Εκεί προσθέθηκε βέβαια και το σημαντικό θέμα των προσφύγων με όλα αυτά που συνεπάγονται. Έχουμε την συμφωνία με την Τουρκία την προσέγγιση της Ιταλικής κυβερνήσεως για τους πρόσφυγες κλπ. Πώς λαμβάνεται υπόψη όλο αυτό στα πλαίσια του προπολογισμού του 2007 εάν προχωρήσουμε με κίνδυνο περικοπών οριζοντίων και με ενδεχόμενη αναθεώρηση ε, κάτι που υπενθύμησε ο εισηγητής. Χρειαζόμαστε πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω κάτι. Το πρόγραμμα Erasmus Plus διότι προσφέρει ενδιαφέροντα εργαλεία όσον αφορά την δράση κλειδί υπαριθμών 2, όπως επανειλημμένα υπογραμμίστηκε από τους άλλους και από τους εκπροσώπους των εκπαιδευτών των νέων, ε, είχαν λιγότερο αποτέλεσμα τα εργαλεία από το προβλεπόμενο και θα ήταν σκόπιμο εδώ να δούμε γιατί, ποια είναι τα αίτια. Πέρα από ότι συμφωνώ με τον κίνδυνο ε, για τον πληρωσμό των λογαριασμών ε, που δεν θέλει εγωιστική προσέγγιση. Η πραγματική αύξηση του προπολογισμού για τη δράση 2, κλειδί δράση 2, θα πρέπει να εξεταστεί λεπτομερώς μόνο το επόμενο έτος 2017. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν η αύξηση για το 2017 που προβλέπεται να έχει αποτέλεσμα που να μην είναι άσχετο, να έχει θετικό αντίκτυπο. Η διαχείριση τέτοιων δράσεων σε επίπεδο αποκεντρωμένο απέδειξε ότι υπάρχουν κάποια όρια όσον αφορά την ανάπτυξη τη καινοτομία και του πειραματισμού, νέε πρακτικέ για να αντιμετωπιστούν πανευρωπαϊκά προβλήματα. Όλα αυτά μπορούν να βελτιστοποιηθούν μόνο μέσω προσεγγίσεω πανευρωπαϊκή, που βέβαια διατρέχει τον κίνδυνο να, καλύψουμε ε, ε, προσπάθειες που γίνονται σε κρατικό επίπεδο. Χρειάζεται συντονισμό. Α πούμε, αναστολή ε, επενδύσεων για την νεολαία στην Ελλάδα έγινε διότι έλειπε εθνικός οργανισμός Άρα ήταν πρόβλημα συντονισμού ε, και το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό. Δεν θα θέλω να αποκλίνω, θα καταλήξω στα συμπεράσματά μου. Το πρόβλημα λοιπόν είναι σημαντικό να ερευνηθεί στο πλαίσιο των ετησίων προϋπολογισμών. Ε, θέλουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο να εφηγραμμίζεται με αυτά που αναδύονται και διαπιστώνουμε ομόφωνα θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βάλουμε και την δράση κλειδί υπαριθμών 2, ούτω ώστε και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το τομέα να έχουμε πανευρωπαϊκά σχέδια. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση, συνάδελφε Σβέρ, έχετε το λόγο. Μα έκανα λάθο, δεν έβγαζα τα γράμματα, έκανα λάθο, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα περισσότερα σχόλια αφορούσαν τη γενική κατάσταση του προπολογισμού. Ε, μιλώ για τον κύριο Γκάιερ τώρα, είναι σοσιαλιστής. δικό του προνόμιο, εγώ δεν είμαι. Αλλά είμαι εξοικειωμένο από την πολιτική στη χώρα μου, από αυτά τα σχόλια. Δεν έχουμε κονδύλια, θέλουμε ένα φιλόδοξο προπολογισμό. Εγώ πάντοτε τρομάζω όταν ακούω να συνδυάζονται αυτές οι δύο λέξεις πολλά άλλα επιπτώσει, τι εργα... δουλεύει, τι δεν δουλεύει, ψηλότεροι φόροι, περισσότερε δαπάνε κτλ. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να οριμάσει ω θεσμικό όργανο, δεν μπορεί να ζητά ε, περισσότερα μετρητά και να είναι οι καλοί που ε, δαπανούν και οι κακοί είναι τα κράτη-μέλη που στέλνουν πίσω του λογαριασμού και τα τιμόλογια. Ε, σίγουρα είναι καλέ οι δαπάνε. Το Erasmus Plus το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι και ξέρετε ότι μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές ως πρόγραμμα, αλλά αυτό σημαίνει επιλογές. Όταν ε, ήμουν πολιτικός στη χώρα μου και ήθελα να δαπανίσω όλα τα χρήματα για τις βιβλιοθήκε, θα έπρεπε να δαπανίσω λιγότερα για λεωφορεία. Αν ήθελα να δώσω περισσότερο για την παιδεία, ε, θα έδινα λιγότερα κάπου αλλού. Και δεν σημαίνει ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν πάντα σε περισσότερες θέσεις εργασίας. Η ομάδα μας λοιπόν η ΣΥΑΡ θέλει δεν θέλει αύξηση μόνο του προπολογισμού, αλλά ισορροπημένο προϋπολογισμό Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και ο υπόλοιπο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να ζει μέσα στις δυνατότητες του. Άρα να ιεραρχήσει τι προτεραιότητε. Ανέφερα μεταξύ των προτεραιοτήτων το Erasmus. Άλλα προγράμματα όμως δεν τα ανέφερα και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε που είναι οι δικέ μου προτεραιότητες Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση, ο συνάδελφε Τόμ, έχετε το λόγο, κύριε Τόμ. Ευχαριστώ. Ομολογώ ότι είχα ετοιμάσει κάτι να το διαβάσω, αλλά μετά σε ένας ευγενικός κύριος που μου λέει ότι δεν έχουμε χρήματα, δεν θα υπάρξουν αυξήσει στον προϋπολογισμό. Οπότε βρίσκομαι σε δύσκολη θέση τώρα. Θέλω να υποστηρίξω αυτό που είπε η Χέλγα Τρούπερ, ότι δηλαδή το Erasmus ε, ΣΥΝ, η ε, Ευρώπη για τους πολίτες, ε, για την Ολή, όλα αυτά είναι προγράμματα πολύ σημαντικά. Είναι ο κραγωνίος λίθος ε, της ε, πολιτικής μας για την νεολαία και σημαντικό αντικείμενο για την Επιτροπή μας. Χρειάζονται αυτά τα προγράμματα και χρήματα. Αν δείτε εδώ αυτά τα έγγραφα ε, που έχω μπροστά μου, που κοστίζουν 3 ευρώ και δεν τα διαβάζει κανείς. Αν τα ξεφορτωθούμε όλα αυτά τα έγγραφα από το γραφείο μας, νομίζω ότι θα εξοικονομήσουν πολλά χρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τα προγράμματα τη Ένωση, για την Όλα. Επίση τυπώνουμε όλα αυτά τα έγγραφα που πρέπει να πηγαίνουμε να τα παίρνουμε και μετά ε, τα ανακυκλώνουν, ε, τα κένα, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να βρούμε πού αλλού θα μπορούσαμε λοιπόν να εξοικονομήσουμε χρήματα και όχι στον πολιτισμό. Είναι λάθος να προσπαθούμε να γλιτώσουμε από εκεί χρήματα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα ζητήσουμε τον εισηγητή να δευτερολογήσει. Έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κρίνει ακόμη την πρόταση για το σχέδιο προπλήσμου 2017. παρόλα αυτά, Θέλω να σας ε, καθησυχάσω ότι τηρούμε τις διατάξεις του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου για τον προπλησμό του 2017 και προβλέπεται μία μικρή αύξηση για το Erasmus Plus. Γύρω στα 200 κάτι εκατομμύρια για το 2017. Βέβαια, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε τις προτεραιότητες για τη χρηματοδότηση ε, του 2017 όταν εγκριθεί. Ο προϋπολογισμός θα έχουν περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά να σας πω ότι ο προϋπολογισμός, μέρος του προϋπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί για τις προτεραιότητες που θα έχουν να κάνουν με την κοινωνική ένταξη και τα εκπαιδευτικά προγράμματα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις τη δήλωση δηλαδή των Παρισίων. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Creative Europe, πάντα στο πλαίσιο του προγραμματισμού μας μέσα στο πολιτές μεσονομικό πλαίσιο, εδώ προβλέπουμε μια ελαφρά αύξηση στο υποπρόγραμμα, στα το... τομεακό υποπρο... στα τομεακά υποπρογράμματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της δανειακής διευκόλυνσης. Θα ξεκινήσει φέτος όπως γνωρίζετε αυτό το πρόγραμμα και θα συνεχιστεί και εντός του 2017. Αυτές είναι οι βασικές μας προτεραιότητες και βέβαια αυτό που περιμένουμε τώρα είναι η πρόταση της Κομισιόν, αλλά σε ό,τι αφορά τα προγράμματα ήδη έχουμε κάποιες σχετικές διατάξεις, οποίες εφαρμόζουμε. Αναφέρεται επίσης και κάποιοι από εσά και θέλω και εγώ να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν προβλήματα, ιδίω στο Erasmus Plus, ό,τι αφορά τι ε, πληρωμών ιδίως το 2014 και το 2015. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα, γιατί δεν υπάρχουν και παρκείς ε, πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να προσθέσω κάποιε σκέψει. Οι συνάδελφοι ήδη κάλυψαν πολύ καλά την όλη προβληματική που αναλύουμε. Εξετίμησα την ειλικρινή γλώσσα. Θέλω και εγώ να είμαι ευθύ αυτά που λέω. Λοιπόν, υπάρχει εμφανής αντίφαση μεταξύ των προσεγγίσεων. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι έχουν πολλά προβλήματα που ζει η Ευρώπη. Η διάσταση της παιδείας και του πολιτισμού των πολιτικών πρέπει να εμφανίζεται πολύ περισσότερο. Όλοι οι επίτροποι και πιο διστακτικοί στα προγράμματά τους προσπαθούν να εντάξουν κάτι που αναφέρεται στο διαπολιτισμικό διάλογο, στην ένταξη, στην ανθρωπιστική κρίση κλπ. Άρα χρειάζονται οι χρηματοδοτούμενες πολιτικές σε αυτό το πεδίο. Ε, πρώτα είναι ένα πολιτικό ζήτημα που τίθεται. Των πολιτικών που θα πρέπει να ετοιμαστούν με πόρους. Τέλεια. Συζητάμε τη μετανάστευση, Φερρυπίν. Δεν θα μπορούσαμε εντός του θέματος μεταναστεύσεως να έχουμε κάποιο ποσό που θα απευθύνεται προς θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ή τον πολιτισμό και διαπολιτισμικά προγράμματα. Παρά να έχουμε προγράμματα όπως η Δημιουργική Ευρώπη που ήδη υποεκτιμάται έναντι των απαιτήσεων που αντιμετωπίζει και να περικόπτουμε πόρους από εκεί για να πάμε σε άλλο τομέα. Όταν μιλάμε για την μεταναστευτική πολιτική, την πολιτική ασφαλείας και εξωτερική πολιτική, εμείς με την πρόταση που έκανε ήδη η κυρία Μογκερίνη για νέα πολιτισμική ευρωπαϊκή διπλωματία. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε αυτές τις προτεραιότητες εντός και των νέων πλαισίων πολιτικών. Είναι θέμα πολιτικής προσεγγίσεως. Δίπλα σε αυτό έχουμε τα προγράμματα. Λαμβάνω υπόψη ότι σύμφωνα με το πολιτές πρόγραμμα έχουμε στο έρασμος για τον επόμενο χρόνο φυσιολογική αύξηση, διότι έτσι είχε προβλεφτεί από τις δόσεις, αλλά μετά στη δράση 2 είναι ότι αντί να αναπτύξουμε εκεί κάποιες πολιτικές καινοτομίες όπως η μαχία για την γνώση, συμπράξεις για την καινοτομία, εμείς προτιμούμε να δώσουμε προτεραιότητα κάνοντας περικοπές από τα προγράμματα και να μην βλέπουμε ότι υπάρχει μία νέα πολιτική για τη μετανάστευση και την ένταξη. Δημιουργική Ευρώπη. Αν δείτε τα τέσσερα βασικά στοιχεία του πολιτισμού θέλουμε να γίνονται η αποδοχή των προγραμμάτων της τάξης του 11%. Άρα οι εμπλεκόμενοι απογοητεύονται. Διότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στον τομέα. Οι νέοι ε, αναμειγνύονται στα πολιτιστικά θέματα. Και υπάρχουν και σχετικές πρωτοβουλίες. Μεγάλος παράγων απασχόλησης και ανάπτυξης ο δημιουργικός αυτός τομέας. Νομίζω ότι και εσύ είσαι ευαίσθητο σε αυτό το θέμα. Ένα άλλο παράδειγμα. Θετικό. Δέχτηκε η Επιτροπή όταν παρήγαγε την έκθεσή του Κοινοβούλιο για την ανθρωπιστική βοήθεια για τα παιδιά στους πρόσφυγες, στην εκπαίδευση των παιδιών στα στρατόπεδα των προσφύγων. Δεν μπορούσαμε να πούμε να δώσουμε πολύ λίγα χρήματα. Δώσαμε μάχη με την Επιτροπή Ανάπτυξης και πετύχαμε 52 εκατομμύρια φέτος να δοθούν παραπάνω για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοηθείας. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να εκφράζουμε περισσότερες πολιτικές. Μετά όσον αφορά το ΕΦΣΥ. Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι. Όσον αφορά το ΕΦΣΥ, ελάχιστα υπάρχουν όσον αφορά τη δυνατότητα επενδύσεων στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας. Κάναμε μια κρόαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, επεξεργαζόμεθα το θέμα, θα εγκρίνουμε το νέο χρηματοδοτικό μέσο για τη Δημιουργική Ευρώπη. Και διαρωτώ στις εκθέσεις του προπολογισμού μήπως θα δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ούτως ώστε αυτό το εργαλείο που είναι σημαντικό να μην δίνει επενδύσεις μόνο για αυτό που είναι ελκυστικό στη συνεργασία με το ιδιωτικό τομέα, αλλά να πάμε πιο πολύ προς την εκπαίδευση να κινηθούμε λίγο. Αυτά, αυτά ήταν οι σκέψεις που είχα και ήθελα να τι μοιραστώ με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συναδελφοί, σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις αυτές που κάνατε και θα προσπαθήσω να απαντήσω στο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Δεν είμαι βέβαιος αν κατάλαβα επακριβώς όλες τις λεπτομέρειες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κάνω ό,τι προσπάθεια μπορώ. Μία πρόταση να πω για τη διαδικασία. Καταρχά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι 25 Μαου θα υποβάλει την πρόταση τη και η πρόταση αυτή θα περάσει πρώτα από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα το επεξεργαστεί την πρόταση αυτή βάσει των κατευθυντήριων γραμμών τη. Θα κάνει κάποιε διαγραφέ, πάντα κάνει και διαγραφέ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τι πληρωμέ γιατί οι δεσμεύσει πληρωμών δεν απασχολούν απαραίτητα, αλλά οι πληρωμέ ε, απασχολούν για να υπάρχουν περιθώρια για τα τα όρια και πάντα μα λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αντίδραση σε έκτακτα περιστατικά. Εμεί με τη σειρά μα θα κοιτάξουμε την πρόταση του Συμβουλίου. Θα κάνουμε αλλαγές και σε πιο πολλές ε, περιπτώσεις ε, εμείς επαναφέρουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά εκεί όπου έχουμε αποφασίσει ότι είναι οι προτεραιότητές μας, υπογραμμίζουμε τα ζητήματα αυτά, αλλά οι κατηγορίες δεν είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες. Δηλαδή, αν τα χρήματα στην κατηγορία 3 που μας απασχολούν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το Erasmus Plus, θα πρέπει να βρούμε χρήματα από την κατηγορία 3, στο εσωτερικό της κατηγορίας 3. Δηλαδή θα πρέπει να μειώσουμε προπολογισμό άλλων προγραμμάτων της κατηγορίας 3. Δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό προκλήθεται. Αυτό δεν το ξέρουν όλες οι αρχές καθορισμού του προπολογισμού και χρειάζεται σε πολλέ περιπτώσει να εξηγήσω για παράδειγμα στο Βερολίνο τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και αν δεν το ξέρουν και στο Βερολίνο, Υποθέτω, φαντάζομαι ότι μπορεί και σε άλλες πρωτεύουσε να μην είναι καλύτερα τα πράγματα, να μην το γνωρίσουν αυτό οι συνάδελφοι. Δεν μπορούμε δηλαδή. Δεν μπορούμε δηλαδή να ε, μειώσουμε προγράμματα του προπολογισμού τα οποία δεν μας αρέσουν για να δώσουμε τα χρήματα αυτά σε, άλλους, ε, σε άλλα προγράμματα. Πάντα τα χρήματα αυτά θα πρέπει να μεταφέρονται εντός μιας κατηγορίας και καταλαβαίνετε λοιπόν το ύφο μου γιατί όταν πηγαίνω στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών καταλαβαίνετε ότι έχουν πολύ διαφορετικές προτεραιότητες για το τι θα πρέπει να γίνει με τα χρήματα της κατηγορίας 3 ε, από ότι εσείς στην δική σας Επιτροπή. Ε, γι' αυτά λοιπόν πρέπει να βρούμε κάποιους λογικούς συμβιβασμούς. Ο συνάδελφος Τσέρ με ρώτησε πώς ε, εξελίσσεται το Erasmus Plus. Όντως, ούτε ήξερα αυτά που μας είπε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν μας το είχε πει η Γενική Διευθύντρια, αλλά από όσον ήξερα, θα, από ό,τι κατάλαβα, θα αυξηθούν κατά 250 εκατομμύρια τα κονδύλια για το Erasmus Plus. Είμαστε λοιπόν πλέον στο 1,73-1,74 δις περίπου. Αυξήσαμε ε, κατά 6,6 εκατομμύρια. Συμβολική αύξηση, γιατί ουσιαστικά δεν έχει οποιοδήποτε μεγάλο αντίκτυπο, γιατί είμαστε φυσικά υπέρμαχοι του Erasmus Plus. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω μα δώσει 250 εκατομμύρια παραπάνω, θα ξεπεράσουμε τα 2 δισεκατομμύρια και είμαι βέβαιο φυσικά το Συμβούλιο θα κάνει περικοπέ. Αλλά να είσαστε βέβαιοι ότι θα επαναφέρει το ποσό αυτό τη αύξηση η Επιτροπή ε, Προπολογισμού του Κοινοβουλίου τι θα γίνει τώρα, σε, πώς θα καταλήξουμε στη συμφωνία με το Συμβούλιο. Αυτό θα κριθεί τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες. Χέλγα, ήσουν συντονίστρια των Πρασίνων στην Επιτροπή Προπολογισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχεις μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη στο θέμα αυτό και φυσικά ο προπολογισμό δεν εμπεριέχει την απαραίτητη ευελιξία. Το ξέρουμε, αλλά και το είπες και εσύ. Αυτό δεν αλλάζει στην ετήσια διαδικασία. Αυτό θα πρέπει να γίνει στην επόμενη αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Θα το ξαναθέσουμε την επόμενη φορά το θέμα. Όταν συζητάμε με εκπροσώπου των κρατών μελών, καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί τουλάχιστον συμφωνούν μαζί μα Τώρα κατά πόσο αυτό θα σημαίνει ότι θα το θυμηθούν την κρίσιμη στιγμή και θα το αλλάξουμε, ε, δεν θα κόβα και το χέρι μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συμφωνούν και λένε, μα γιατί δεν υπάρχει παραπάνω ευελιξία. Πάντα είμαστε σε επαφή με τους ε, από τα Υπουργεία Οικονομικών. Τώρα θα γίνει την ώρα τη κρίση δεν ξέρουμε. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο εισαγάγαμε κάποια εργαλεία μετά από μεγάλη προσπάθεια του Κοινοβουλίου που εισαγάγουν κάποια ευελιξία παρά την αντίσταση των κρατών μελών. Και αν δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα ευελιξίας, ε, το περασμένο έτος ε, θα μας είχε τεινάξει στον αέρα λόγω της προσφυγικής κρίσης. Δίκιο λοιπόν είχαμε. Αποδείχθηκε αυτό. Και θα συνεχίσουμε να το υπογραμμίζουμε αυτό. Ύστερα, μίλησε και για τη διαδικασία υποβολή αιτήσεων. Αυτό ασφαλώ στον προπολογισμό. Θα το δείξουμε όπω και στην πολιτική διακήρυξη. Δεν το θίγουμε ιδιαίτερα στην ε, αναθεώρηση. Εγώ ήμουν υπεύθυνο για την πολιτική ελέγχου του προπολογισμού και αυτό αποτελεί σημαντική υπότεξη για τους συναδέλφους της Επιτροπής. Κοιτάξτε τι κάνουν οι εθνικές, τα εθνικά ιδρύματα, οι εθνικές υπηρεσίες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος κατά πόσον ε, το γραφειοκρατικό άχθος το οποίο πάντα επικρίνεται προέρχεται από εμά, από, από απαιτήσει που θέσει το Κοινοβούλιο ή από προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό είναι μια δυνατότητα, αλλά εγώ τι έχω δει από τον τομέα του ελέγχου του προπολογισμού. Ότι τα εθνικά, οι εθνικές υπηρεσίες ενδεχομένως να περιπλέκουν τη διαδικασία υποβολής απτήσεων. Οι εθνικές υπηρεσίες. Αυτό το ακούω ως καταγγελία συχνά. Και σίγουρα αξίζει τον κόπο τουλάχιστον στη Γερμανία, να ελέγξουμε κατά πόσον η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το Erasmus Plus επιβάλλει επιπλέον προδιαγραφές σε μια ευρωπαϊκή ρύθμιση, επιβάλλοντας δηλαδή εθνικές υποχρεώσεις. Άρα, εντάξει, Κάποιε φορές ε, τα περιπλέκει πράγματα και το ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά όχι μόνο το ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν φταίνουν μόνο οι Βρυξέλλε. Ύστερα, στο επόμενο θέμα, Όντω. Ε, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και λίγο πιο περίπλοκα. Δεν θέλουμε απλά πιο πολλά κονδύλια, πιο πολλά χρήματα. σε κάποιε περιπτώσει υπάρχουν κάποια επιχειρήματα, γιατί σε κάποιε περιπτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει νέε αρμοδιότητες και η χρηματοδότηση αυτών των νέων αρμοδιοτήτων δεν είναι αντίστοιχη. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε να το σκεφτόμαστε αυτό. Κατά πόσον η Frontex με το ίδιο όνομα μπορεί να αναλάβει συντονισμό κάποιων άλλων υπηρεσιών σε πιο πολύ λειτουργικό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε τελική ανάλυση τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενισχυθούν οι εργασίες απλά. Μπορούμε να βάλουμε στοίχημα κατά πόσο λέει η θέση του Συμβουλίου η οποία θα προκύψει. Θα το αποτυπώνει αυτό. Θα αποτυπώνει αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει ω αύξηση στην κατηγορία 3. Στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποτυπώνεται. Αλλά αν θέλουμε η προστασία των συνόρων να καταστεί πιο πολύ ευρωπαϊκό ζήτημα, τι γίνεται με τι πληρωμέ από πλευρά ε, Συμβουλίου. Και αν γίνεται από το από ευρωπαϊκή πλευρά θα πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο, αντίστοιχο από εθνική ε, πλευρά. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει αρμοδιότητε. Ε, το εθνικό επίπεδο αποσυμφορείται κάπω, όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, και δεν μπορούμε να πούμε ότι το Κοινοβούλιο πάντα επιμένει για πιο πολλά χρήματα. Όχι. Ε, λυπάμαι. Αυτό που, στο οποίο επιμένουμε είναι ότι για νέε αρμοδιότητε, για νέε ευθύνε πρέπει να υπάρχει και μια χρηματοδότηση. Το γνωρίζω λοιπόν το επιχείρημα αυτό. Αλλά για να σας παρηγορήσω και στην Βρετανική συζήτηση, να σας πω το εξή. Κάντε λίγο μια προσπάθεια, κάντε ένα κόπο και κοιτάξτε τις ειδικές εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. που κάνουν τεγματοληψίες σε διάφορες χώρες και τελικά, ας το θέσω έτσι. το Ηνωμένο Βασίλειο την γλιτώνει φτηνά σε ό,τι αφορά τις ειδικέ εκθέσεις ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, για παράδειγμα, της υπαίθρου. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να οθήσει την εθνική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας να κοιτάξει τι γίνεται με τον έλεγχο τον εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου για τις ε, δαπάνες των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Αν ε, λοιπόν επικρίνεται τα ευρωπαϊκά έξοδα, Κοιτάξτε τι γίνεται και στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί έχετε με πολλή δουλειά μπροστά σας. Και να κλείσω λέγοντας το εξή. Να πω και το εξή προς τους συναδέλφους. Δεν θέλω να είμαι άδικος και πολιτικά Κατανοώ αυτά που λέτε για την πρόθεση της πολιτικής για τα πολιτισμικά, αλλά με τα χρήματα που ξοδεύουμε για την προσφυγική κρίση, ε, χρηματοδοτούμε και πρωτοβουλίες της UNICEF. Για παράδειγμα για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα και θα πρέπει φυσικά από πλευρά τη Επιτροπή σα να συμπεριλάβουμε και προτάσει επί του περιεχομένου. Έχουμε το εξή πρόβλημα, ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τον προπολογισμό όσο έχει, τι κατηγορίε όσο έχουν, τα όρια όσο έχουν. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Γιατί η παράθεση για τον προπολογισμό συνήθως έχει να κάνει με ποσά τα οποία είναι 3 έως 5% πολύ πιο μεγάλα άλματα δεν μπορούμε να κάνουμε και να είστε βέβαιοι ότι τα προγράμματα τα οποία θίξατε θέλω να τα εξετάσω όλος ιδιαίτερος ότι με απασχολούν όλος ιδιαίτερος ως εισηγητής Έχετε και την έκθεσή σα, την γνωμοτότησή σα στην Επιτροπή Προπολογισμού για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε λοιπόν αυτά και εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την ειλικρίνεια τη απαντήσεω. Σίγουρα Κοιτάξτε, ο συνάδελφο Τρογεύσκη είχε ένα πρόβλημα, άλλη μέρα θα είναι παρόν, να διευκρινίσω κάτι. Εμεί δεν θέλουμε να διερευνήσουμε τι επενδύσει, τις αρμοδιότητες. Ξέρουμε ποια είναι τα όρια. Είναι σημαντικό στα πλαίσια των άλλων πολιτικών να αυξηθεί η προσοχή στο περιεχόμενο που είναι ο πολιτισμικός και εκπαιδευτικός στόχος. Λοιπόν, δώσαμε μάχη για να αυξηθεί η ποσόστοση στα πλαίσια ανθρωπιστικής βοήθειας για την εκπαίδευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ζητάμε παραπάνω χρήματα. Ζητάμε να, η ανθρωπιστική βοήθεια να μην είναι μόνο το 2%. Δεν θέλουμε να διαχειριστούμε εμεί το κεφάλαιο, την κατηγορία αυτή, αυτό είναι σαφές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί ελπίζω να κάνουμε έξοχη δουλειά. Σας εύχομαι καλή δουλειά, διότι το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με αυτό ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση. Παρακαλώ τους συντονιστές να παραμείνουν, αν έχουν την καλοσύνη συντονιστές, και οι άλλοι όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται στη συνεδρίαση των συντονιστών παρακαλώ να αποχωρήσετε και ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας.